Καλημέρα συνάδελφοι, συνάδελφοι της εργασίας της 9.30 έχουμε συνάντηση με τον Επίτροπο υπεύθυνο για θέματα περιβάλλοντος, τον κύριο Ποτότσνικ και δεν μπορούμε να, να επιτρέψουμε καθυστερήσεις. Έχουμε δύο σημεία που θα πρέπει να εξετάσουμε. Δεν υπάρχει πυκνή παρουσία των συναδέλφων. Εγώ θα ξεκινούσα λοιπόν το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης να σας δώσω ε, μια παρουσίαση των αποφάσεων που έλαβαν αυτές το βράδυ οι συντονιστές ε, κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως τους που συνεδρίασαν από 5.30 μέχρι 6.30. Τα σημεία της ημερής διάταξης συνεδριάσεως ήταν 6 επί του πρώτου σημείου. Οι συντονιστές ε, συζήτησαν κάποια κριτήρια για τον καθορισμό των εισηγητών ε, και έπρεπε να καθοριστούν συγγητή για τρία έγγραφα που θα εξεταστούν από την Επιτροπή μας, πιο συγκεκριμένα ε, η έκθεση για την ετήσια έκθεση του 2011, οι δραστηριότητε της Επιτροπής μας, γνωμοδότηση για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μια γνωμοδότηση που θα πρέπει να ανατεθεί ακόμα όσον αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά το σύστημα για τα ύδατα. Οι συντονιστές επ' θα αποφασίσουν ε, στην επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Μετά εξετάσαμε τη διαδικασία για την καλύτερη διαχείριση των αναφορών ε, των διαφόρων ε, καταγγελιών που δεχόμαστε από τους πολίτες πάνω που πριν από 6 μήνες, πάνω από 6 μήνες εκεί στη δικασία και αποφάσισαν συντονιστές χτες να επικαιροποιηθεί όλος ο προβληματισμός ε, στην επόμενη συνεδρίαση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τελικά το πρότυπο που η γραμματεία ετοιμάσε του εγγράφου που δυστυχώς χθες μόλις το απόγευμα δόθηκε και θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Όσον αφορά το σεμινάριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα που έλαβε χώρα στις 6 Οκτωβρίου, ε, οι συντονιστές χθες το βράδυ αποφάσισαν να προωθήσουν ανοιχτή συζήτηση στην Επιτροπή, δηλαδή να, να προβλέψουμε κάποιο χρόνο σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής αφού έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να να συλλέξει τις ομιλίες όλων εκείνων των ομιλητών που μίλησαν στο σεμινάριο και πάνω σε αυτά που είπαν να είναι πιο περιστατωμένη συζήτηση. Θεωρεί, ε, είδαμε επίσης ότι διεξήχθη μια ανάλογη συζήτηση διοργανωθής από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και συνάδελφοι πάνω σε αυτό πρότειναν αυτή η ανοιχτή συζήτηση να λάβει χώρα σε μια μεικτή επιτροπή, ε, Επιτροπής Αναφορών, Επιτροπής Δημοσίων ε, Ελευθεριών. Αυτή η διαδικασία θα λάβει χώρα τους επόμενους μήνες και θα αναπτυχθεί. Όσον αφορά την πρωτοβουλία των, ε, πρωτοβουλίας των πολιτών, τις περασμένες εβδομάδες, μάλιστα τους προηγούμενους μήνες, μα ενημέρωσε η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη μία αντιστοιχεία των ε, πληροφοριών που χορηγήθηκαν από την Επιτροπή ΑΦΚΟ ε, όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και τις εγκρίσεις του κανονισμού για την πρωτοβουλία των πολιτών. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Επιτροπή μας, η Επιτροπή των Αναφορών, θα έπρεπε να διαδραματίσει ένα ρόλο στη φάση που, θα προηγηθεί της Έναρξη τη νομοθετική διαδικασία πρώτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όσον αφορά τις προτάσεις που πληρούν ω προποθέσει ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν ω πρωτοβουλίε ε, των πολιτών. Η ΑΦΚΟ στην ε, πρότασή της με τις ε, τροπολογίες που υπευλήθησαν όσον αφορά την εμπλοκή της Επιτροπής Αναφορών την αναβάλει σε επόμενη φάση και είναι ένα ενδεχόμενο όπου μια πρόταση που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του ώστε να θεωρηθεί ε, ως πρωτοβουλία των πολιτών μεταφέρεται στην, ε, θεωρείται αναφορά και μεταφέρεται στην Επιτροπή μας. Αυτό δεν προβλεπόταν συμφωνίες μας, δεν ήταν αυτό που η Επιτροπή μας είχε συζητήσει. Συνεπώς οι συντονιστές αποφάσισαν να διεκδικήσουν σε πολιτικό επίπεδο ο καθένας στρεφόμενος προς το πολιτικό του φορέα να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν κατά τη φάση των συζητήσεων των λόγω κανονισμού που μετά ενεκρίθη πάρα πολύ γρήγορα. Άρα να υπάρξει επιμονή όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού και πιο συγκεκριμένα του άρθρου εκείνου που προβλέπει ποιε είναι οι αρμοδιότητες επιτροπή των Αναφορών εισάγοντας και αυτή την φάση της διαδικασίας των, της πρωτοβουλίας των πολιτών. Όσον αφορά το παλιό θέμα του νόμου ε, λέει δε Κώστας, ε, οι συντονιστές επιβεβαίωσαν την όλη ιδέα του να μην τοφοδοτηθεί υπερβολικά μια συζήτηση που θα συμπεριλαμβάνει υπερβολικούς όρους και να παραμείνει ε, χαμηλός ο τόνος ε, επί θέματος που απασχολεί επί σειρά ετών αυτή την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Υπογραμμίστηκαν επίσης και οι ανάγκες να μην, να μην πέσουν στο κενό οι διάφορες πρωτοβουλίε των πολιτών, να δοθεί συνέχεια και να καταβληθούν προσπάθειες για την εξέβρεση συγκεκριμένη λύσεως. Για να γίνει αυτό και για να μην εργαστούμε υπό την πίεση την κατανοητή των πολιτών οι συντονιστές θέλησαν να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας και θα καθοριστούν τα μέλη της επόμενης εβδομάδας και η ομάδα εργασίας αυτή θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση των ενδεχόμενων λύσεων και διαδρομών που ακολουθηθούν και θα προθύνει τελικά στην Επιτροπή μας την πρωτοβουλία που θα πρέπει να υιοθετηθεί. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε να ανακοινωθεί να κοινοποιηθεί όταν σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας το πού βρίσκεται αυτό το θέμα που είναι άκρως ευαίσθητο στην Επιτροπή μας, στο Κοινοβούλιο ούτως ώστε η νέα κυβέρνηση να μπορεί να ανακοινώσει τη θέση της και αυτό να μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε ενδεχόμενε δυνατότητες ε, νέων συνεργασιών με τις Ισπανικές αρχές. Εγκρίθηκε μετά η μερίσια διάταξη που προτάθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Και τέλος, ακούστηκαν διάφορες ενδείξεις και συζητήθηκε μια ανακοίνωση που αφορά τη δημιουργία, κατασκευή μιας γέφυρας σε περιοχή Natura 2000 επεστήθη η προσοχή των συναδέλφων άνευ συζητήσεω και επεσήμανα το αίτημα τη του κυρία Αντζελίλη να καθοριστεί υπεύθυνο στην προστασία δικαι... της κυρίας Αντζελίλη μάλλον για τα δικαιώματα των ανηλίκων. Χάρη στην παρέμβαση τη κυρίας Αντζελίλη δημιουργήθηκε μια συμβουλευτική επιτροπή για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε επιτροπή που θα έχει την αρμοδιότητα εντό τη επιτροπή αυτή να προωθεί και να υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες εκείνες που έχουν σαν στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Δύο υποψηφιότητες ακούστηκαν. Η τελική απόφαση όσον αφορά αυτές τις υποψηφιότητες ε, θα ληφθεί τις επόμενες εβδομάδες. Δεν υπάρχουν άλλες αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές. Αν οι συνάδελφοι δεν έχουν αντιρρήσει σχόλια, εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο προβλέπει την έγκριση της έκθεσης όσον αφορά την επίσκεψη στη Βουλγαρία και πριν από αυτό θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Άουκεν έχοντας υπογραμμίσει πρώτα ότι είχαμε έτοιμα μερικής αλλαγής τροποποίησης από πλευράς της συναδέλφου Λεντετσέβα που υποστηρίχθηκε από τη συνάδελφο Άουκεν η οποία θα μας εξηγήσει αυτές τις μικρές αλλαγές και παρεμβάσεις και θα σας παρουσιάσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε την ε, αναφορά και πρότεινε η κυρία από τη Βουλγαρία μια σειρά τροπολογιών ούτως ώστε να υπάρξει κάποια διόρθωση των πραγματικών περιστατικών. Ε, ο Γκουίντε Παντοβρή, αν θέλει και ε, δεν ξέρω ε, ε, αν, μπορεί να συμφωνήσει. Για μένα είναι εντάξει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά κάποια στοιχεία εδώ για την Επιτροπή μας. Πρώτα-πρώτα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά ελπίζω ότι πρόκειται να εξασφαλίσουμε παρουσία μεγαλύτερη των μελών. Ε, τέλος πάντων πρόκειται για μια επίσημη αντιπροσωπεία και έτσι προσπαθήσαμε να έχουμε ε, δύο από τη Βουλγαρία, τελικά μόνο ένα εμφανίστηκε και δηλαδή να μπορούμε να προβληθούμε περισσότερο. Και είχα, είχαν ακόμα οργανώσει και κάποιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, οπότε έτσι πρόβαλαν το θέμα τους και τελικά ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι όταν επισκέφθηκε τη χώρα έγιναν τα ίδια. Οπότε, πώ να το πω, έτσι να το πω διπλωματικά μας έφερε σε αμηχανία. So you have the feeling that you are dealing with a... Οπότε προσπαθούμε να δούμε τι προσπάθειες καταβάλει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη της οικονομίας, της βιομηχανίας ειδικότερα και προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται με αυτές τις κοινοπραξίες, τις joint ventures, είναι θεωρητικά πάρα πολύ καλή ιδέα, όμως θεωρητικά, γιατί στην πράξη αυτό που το οποίο συμβαίνει είναι άφατη διαφθορά. είναι στρεβλώνται τιμές κλπ. λοιπά Πάρα πολύ ενισχυτικά όλα αυτά. Ε, τελικά το κοινωνικό δίκαιο εκεί πέρα εκλαμβάνεται ως σύσταση στην καλύτερη περίπτωση και τελικά κατησχύει το εθνικό δίκαιο. Έτσι. Αντιλαμβάνω τα πράγματα, τουλάχιστον εκτός σόφιας. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς τελικά θα γίνει σεβαστό το κοινωνικό δίκαιο. Τώρα που θα συναντήσουμε τον Ποτότσι, νομίζω θα πρέπει να το τονίσουμε όλα αυτά. Έχουμε ένα σωρό δεν θα πρέπει να το πούμε. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σοβαρά το ρόλο της. Και να κάνει κάτι όταν έχουμε μια κατάφορη παραβίαση του γενικού δικαίου. Γιατί έτσι γίνεται. Μα είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιε δραστηριότητε που να πιέσονται μέσα σε περιοχή του Natura 2000. Αυτό γίνεται σε μια σειρά τόπων. Δεν του νοιάζει. Στα βουνά αυτά είναι υπέροχα εκεί που έχουν τα, σκι. Ακόμα και συναυλίες ρόκαν, είναι τόσο όμορφα, έχουν αυτά τα, τις βίλες εκεί πάνω στο βουνό στη Αλλά έβρεχε, σχεδόν χιόνιζε και δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί. Πάρα πολύ δύσβατη περιοχή. Και εκεί, πάνω πάνω στο βουνό, ξαφνικά βλέπουμε ένα σπίτι. Τι είναι αυτό λέμε. Αυτό ήταν αυθαίρετο, πολύ αυθαίρετο. Και όμως, κοίτας, και μας είπαν ότι είναι τουριστικό περίπτερο. Υπέροχο. Είναι υπέροχο μέρος, ναι. Όλα αυτά τα κάνανε για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια λεφτά, βέβαια. για την μεταφορά, για ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να χτίζουν εκεί που έχει τα δέντρα, να τα κόβουν και Sure, that we don't have conflicting rules in the, uh, uh, in the EU system. I think we should. Και έτσι πήραν τα κονδύλια της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Για να δούμε μόνος για όλες τις περιπτώσεις. Να μην είναι πρόφαση η ΚΑΠ και να κόβουν τα δέντρα σε τέτοια ωραία μέρη. Πάντως το θετικό ήταν ότι οι αναφερόμενοι ήταν πάρα πολύ καταρτισμένοι. ειδικοί, ο κόσμος, έχει παραγωγές δυνατότητες. Είναι καταρτισμένοι λοιπόν και επομένω είναι τεκμηριωμένε οι αναφορέ. Άρα και εμεί θα πρέπει αυτόν τον να γνωρίσουμε του αναφερομένου για όλα αυτά τα οποία μας μαθαίνουν. Γιατί αυτά τα βουνά τη Ρίλα είναι ευρωπαϊκή κληρονομιά, όχι βουλγαρική. Είναι ευρωπαϊκό αυτό το υπέροχο μέρος. Άρα θα πρέπει να το φροντίσουμε. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πιο διπλωματικά διατυπωμένα. I could I will finish by saying that again this uh, ongoing. Μπορείτε να το δείτε σε αυτέ τις συναντήσεις που έχουν γίνει ε, και με στενή συνεργασία με τις αρχές της χώρας αλλά και σε συνεργασία με τους ε, εργολάβους σε εκείνες συναντήσεις διαπιστώσαμε ότι ήταν υποψίαστη για την ύπαρξη του προβλήματος. Ούτε καν προσπαθούν να, να ε, κρύψουν αυτή τη συμπερνία. Να, ποια είναι η πιο σκληρή, η πιο δύσκολη πρόφαση, ε, πρόκληση που έχουμε για το μέλλον σε σχέση με την Βουλγαρία. Και επομένως θα πρέπει να την πλαισιώσουμε την κοινωνία των πολιτών για το αξίζουν. Αυτό γιατί ακριβώ είχαμε αυτή την τόσο θετική εικόνα τότε που πήγαμε στα βουνά τη Ρίλα. Υπάρχει εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να πάρει το λόγο. Α Ας μιλήσει πρώτα ο κύριος Κάσμαν και μετά θα δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Μπουστινάρου. Um, thank, thank you, um, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώ ήρθατε με ιδιαίτερα την έκθεση αυτή. Αναφέρθηκε ότι ο Επίτροπο Ποτόσνικ θα έρθει εδώ συντόμω και ελπίζω να σχολιάσει όχι πάνω στην έκθεση αυτή, αλλά πάνω στα θέματα που αφορά αυτή η έκθεση και που έθιξε η κυρία Άουκεν. Χαιρετίζουμε την ε, διερευνητική επιστολή που έγινε ε, από την Επιτροπή Αναφορών γιατί αυτό μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε μια δική μας κρίση. Υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις σε διάφορα σημεία και καλός αντίκτυπος πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Άοκεν. Ευχαριστώ. Κολέγα Μπουστινάρου. Ο συνάδελφος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τη συνάδελφο Μάργα Άοκεν για την έκθεσή της, την παρουσίασή της. Και για τις τροπολογίες σε σχέση με τις απόψεις των ε, μελών της Επιτροπής, αλλά και των άλλων εμπλεκομένων σε εκείνη την αποστολή. Πάρα πολύ ακριβής ήταν η περιγραφή των όσων γίνονται στη Βουλγαρία. Το θέμα να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες ερευνητικές ε, αποστολές. Θεωρούμε ότι αυτή η διαβούλευση μεταξύ των αρχών και του κόσμου ακόμα είναι ανεπαρκής. Τυπική, πολύ. Απλώς για να λένε ότι την κάνανε. Δεν είναι ευθεντική πραγματική διαβούλευση. Ούτε βοηθάει. Ούτως ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος. Και επομένως δεν συμμετέχει ο κόσμο ούτε μη τι οργανώσει. Επίση, έχουμε εδώ πέρα έλλειψη διαλόγου ή τέλο πάντων επαρκή του διάλογο μεταξύ των αρχών και ε, των ενδιαφερομένων ε, ε, πόλεων και κοινοτήτων. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στη Σόφια αλλά και αλλού. Τρίτον, το οποίο ήδη το ανέφερε η, η Μαργαρίτα, είναι το ότι, πώς να το πω, όσο πιο πραγματικά γίνεται, ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολες, πάρα πολύ ε, περίεργες σχέσεις μεταξύ των ε, αρχών και των επενδυτών. Όλοι μαζί καταπατούν πολύ βασικές αρχές της κοινωνικής νομοθεσίας. Οπότε έχουμε και αυτή την ενημέρωση από το Υπουργείο, από τις τοπικές αρχές που έγινε όταν σκεφτήκαμε το Σαπαρέβο Μπάνια, μας είπαν όλα καλά, όλα στρογγυλά, αλλά στην πραγματικότητα ε, πρόκειτο για τελείως διαφορετική πραγματικότητα όπως επί το που είδαμε. Επομένως, είναι αναξιόπιστες οι πληροφορίες που μας δίνουν οι επίσημες αρχές. Άρα θα πρέπει σε τέτοιες περίεργε ευαίσθητε, δύσκολε περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πηγαίνει επί τόπου για να βλέπει και να διαπιστώνει ποια είναι η πραγματικότητα. Ακριβώ όπως έγινε και με εκείνα τα αιωλικά πάρκα. Έτσι. Να μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση, πλήρη εικόνα για το τι ισχύει. Τέλο. Κατόπιν τη επίσκεψη. αυτό, αυτό είναι το τελευταίο που θα σα πω τι θα γίνει την ε, επαύριο. Πρόκειται να βελτιώσουν τίποτα ή η κατάσταση. Several other fact-finding visits. This are uh, all my points. Thank you. Αυτό θα πρέπει να γίνει επομένω, αυτό θα λάβουμε υπόψη στην επόμενη ερευνητική πραγμάτων επιτροπή που θα πάει εκεί. Ε, Ευχαριστώ συνάδελφε Μποστινάρου. Καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Πατότσνικ που ζήτησε, έχει την καλοσύνη να αποδεχτεί την πρόσκλησή μα για μια ακρόαση θα του δώσουμε το χρόνο να α, τακτοποιηθεί και έτσι θα τον χαιρετήσουμε όπως το αξίζει. Αυτή η ακρόαση ήταν διακαής πόθος των συναδέλφων. Διότι καθημερινά η Επιτροπή μας εξετάζει θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Οι περισσότερες αναφορές που απευθύνονται στην Επιτροπή μας αφορούν το περιβάλλον, Καλωσορίζω τον Επίτροπο Ποτότσνικ. Τον ευχαριστώ που απεδέχθη την πρόσκλησή μας. Όπως έλεγα στην εισαγωγή μου, το περιβαλλοντικό ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο είναι εκείνο που αντιμετωπίζεται στην πλειοψηφία των ε, αναφορών που υποβάλλονται στην Επιτροπή μας. Περίπου 1.200 αναφορές που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή μας για περιβαλλοντικά θέματα. Από αυτές 460 ε, είναι ανοιχτές. Οι περισσότερες αναφορές, οι ανοιχτές, αφορούν οι καζόμενες παραβιάσεις οδηγιών περιβαλλοντικού περιεχομένου, οδηγιών ε, Natura 2000, οδηγιών για τα απόβλητα. Αυτά είναι τα θέματα που καταγγέλλονται περισσότερο από τους πολίτες. Τα θέματα αφορούν περισσότερο την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αυτά είναι τα κράτη-μέλη από τα οποία πιο συχνά μάλλον φτάνουν τέτοιες υποθέσεις ε, διαμαρτυριών καταγγελιών από πλευράς πολιτών. Οι ανησυχίες των πολιτών που απευθύνονται προς εμάς αφορούν την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου που στις περισσότερες ε, περιπτώσεις θεωρείται σαν μη ενδεδειγμένη ή σαν ανεπαρκή σε περίπτωση προγραμμάτων που αφορούν υποδομές ή στον ευρύτερο τομέα των, αποβλήτων. Όσον αφορά αυτού του είδους τις καταγγελίες, οι πολίτες ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες να συμφωνήσουν με τις προβλέψεις της νομοθεσίας που δέχεται την παρέμβαση από πλευράς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπροσωπείτε εσείς, αλλά εν γέννη παρέμβαση από πλευράς των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για την επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας μόνο όταν τελικά έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Κάθε φορά που γίνεται μια καταγγελία που προηγείται της υλοποίησεως ενός έργου που παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι υπηρεσίες, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα της, διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον μας επισημαίνουν ότι δυνατή μια παρέμβαση διότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να αναλυφθεί μόνο μετά την ε, πραγματοποίηση της βλάβης που καταγγέλουν, τις εικαζόμες που καταγγέλουν οι πολίτες. Η Επιτροπή μας, ε, η Γενική Διεύθυνση μας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπροσωπείτε εσείς κύριε Ποτότσνικ, συνεργάζεται μαζί μας, αξίζει αυτή η συνεργασία με την Επιτροπή μας, πέρα από την καλή βούληση που κάθε ένας διαθέτει σε αυτό που κάνει, υπάρχουν όμως και δυσκολίες όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Αυτή η ακρόαση λοιπόν ε, έχει σαν στόχο σύμφωνα την πρόθεσή μας όχι μόνο να διερευνήσουμε ή δυνατόν συγκεκριμένων λύσεων σε πραγματικά προβλήματα που ε, τίθεται στην προσοχή μας πάντα προσπαθώντας να προωθήσουμε μια υγιή συνεργασία σεβόμενη τα δικαιώματα των πολιτών αλλά θέλουμε επίσης να βρούμε τρόπους, ενδεχόμενους τρόπους, για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, ε, να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι αληθεύει ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι εκείνη που είναι καθήλυν αρμόδια πριν από όλες τις άλλες για θέματα περιβαλλοντικά όμως εξίσου αληθεύει για τους λόγους που ανέφερα και για τους αριθμούς που προανέφερα η Επιτροπή μας είναι ο κόδων του κινδύνου που δεν μπορεί να αγνοείται και θα πρέπει να δώσουμε κάποια συνέχεια ούτω ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά θετικοί όσον αφορά τις προτάσεις που θα κάνουμε για θέσπιση νέας κοινοτικής νομοθεσίας ή για την βελτίωση της αλόγω νομοθεσίας, της υφισταμένης νομοθεσίας. Ε, κύριε Επίτροπε, πιο συγκεκριμένα, έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες μέσω επιτοπίων αποστολών για θέματα επί των οποίων έχουμε λάβει πάνω από ένα αίτημα των πολιτών. Και επί μακρόν η Επιτροπή μας έχει κληθεί να δώσει απαντήσεις. Εγώ θα επεσήμενα μεταξύ αυτών των καταγγελιών όχι μόνο το πιο επίγον ζήτημα του σεβασμού των κανονισμών για τα απόβλητα διότι το Δεκέμβριο έχουμε προγραμματίσει την εξέταση στην Σύνοδο του Στασβούργου, στην Ολομέλεια του Στασβούργου, συζήτηση εκθέσεως που αποφασίσαμε να υποβάλουμε στην Ολομέλεια, που ξεκινώντας από τις πολυάριθμες αναφορές που υπευλήθησαν στην Επιτροπή μας, μας οδήγησε να σας προτείνουμε, να προτείνουμε στη Γενική Διάθεση Περιβάλλοντος διορθωτικές παρεμβάσεις, που είναι καρπός εμπειρίας που ορίμασε μέσω καταγγελιών που συζητήθηκαν και εξετάστηκαν και παληθεύτηκαν επί τόπου. Όπως στην καταγγελία που αφορά τα απόβλητα στην καμπανία. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα αίτημα επικαιροποίηση, ενημέρωσης, γιατί όσον αφορά αυτό το γεγονός, αυτό το πρόβλημα, έχει αναλυφθεί δέσμευση από αυτή την Επιτροπή να επιστρέψει στην Ιταλία. Έχει προγραμματιστεί μια επιστολή στην Ιταλία, επιστροφή στην Ιταλία για να δούμε πόσο έχει προχωρήσει όλη η δουλειά. Αλλά μετά ε, ε άλλη επιστολή όχλης από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά αυτή την επιστολή δεν έχουμε περισσότερα νέα και πληροφορίες όσον αφορά την αντίδραση. Και κάτι άλλο που θα έπρεπε να προσέξετε ή δυνατόν και θα θέλαμε και κάποιες πληροφορίες είναι η οδηγία για τα πτηνά και η οδηγία για τους βιοτόπους, habitat. Όσον αφορά αυτό το θέμα, πολύ συχνά η Επιτροπή μας καλείται να συζητήσει και να το εξετάσει έχουν επισημανθεί ελλειπείς εφαρμογές της νομοθεσίας στη Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία και σε άλλες χώρες της Ενώσεως. Έχουν υποβληθεί συγκεκριμένα αιτήματα, κάποια συγκεκριμένα αιτήματα μέσω των αναφορών που έχουν υποβληθεί ή που διατυπώνονται προς την Επιτροπή. Εγώ επ' αυτών των δύο ζητημάτων των συγκεκριμένων θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε κάποια απάντηση, ούτως ώστε να μας επιτρέψετε να προχωρήσουμε με θετικό τρόπο στις εργασίες μας και να μην αφήσουμε αναπάντητες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε έναντι των Ευρωπαίων πολιτών, έναντι των οποίων είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, θα σας δώσω το λόγο τώρα. το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, μέλη τη Επιτροπή, είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθα σήμερα εδώ να σα μιλήσω και ουσιαστικά για πρώτη φορά και γι' αυτό και θέλω να σα ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, τόσο ώστε να μπορέσω να μιλήσω προ την Επιτροπή σα και διότι όπω θα γνωρίζετε, ε, για μένα ε, η υπόθεση τη ε, υλοποίηση των όσων λέμε είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό, οπότε μπορείτε να με θεωρείτε ως έναν πάρα πολύ σημαντικό σύμμαχο και Βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται με, με όλε αυτέ τι ε, επιτροπέ που αφορούν τι παραβιάσει του κοινωνικού δικαίου όσον αφορά το περιβάλλον. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ε, μια αξιολόγηση όσον αφορά το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, αυτό το οποίο, ε, το οποίο δείχνει το πόσο σημαντική πρόκληση θέλουμε το περιβάλλον και γι' αυτό και εμεί θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερο για να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι προβλέπεται υλοποιείται. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται όσον αφορά την ε, νομοθεσία, όπω η νομοθεσία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το πώ θα υλοποιηθούν όλε αυτέ τι διαδικασίες, πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Διότι έχει σημασία η εφαρμογή μια που αφορά την ευημερία, αφορά το, το, ε, την ποιότητα ζωή τελικά των Ευρωπαίων. 20 με 50% των Ευρωπαίων ζουν σε περιοχέ όπου έχουμε ποιότητα της ατμόσφαιρας που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ποιότητα που επιδέχεται βελτίωση. Επομένω, με αυτή την έκθεση είπαμε ότι το κόστος της μη εφαρμογή η νομοθεσία είναι 50 δις ετησίω. Οπότε έχουμε πάρα πολύ σημαντικά κέρδη για την οικονομία. Αν υπάρχει στήριξη των όσων προβλέπει η νομοθεσία, θεωρείται ότι αυτό θα φέρει 600.000 θέσει εργασία και 67 δις θα εξοικονομήσουμε σε σχέση με το εάν δεν εφαρμόζεται η κειμένη νομοθεσία. Άρα μπορούμε σίγουρα να ωφεληθούμε από την, την, το, το, να πιάσει τόπο η δουλειά σας τέλος πάντων, γι' αυτό και την σεβόμαστε το έργο και το έργο σας. Οπότε όπως είπατε ε, είμαι θα, φυσικό το τρόπο σύμμαχη και άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η δουλειά μας και γι' αυτό ε, προς την κυρία Ματσόνη δεν μπορώ παρά να νιώθω ευγνωμοσύνη ε, και ακριβώς διότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τι επαφέ μου με του εμπλεκομένου τον ε, Ιούνιο. Και εμεί πάντω έχουμε το ρόλο του φύλακα των συνδικών. Εσεί πάντω δίνετε την πολιτική διάσταση σε αυτήν όλη την υπόθεση για την παρακολούθηση τη εφαρμογή. Και τελικά η πολιτική διάσταση του πράγματο φαίνεται σε πολλά σημεία. Ε, γιατί προερχόμαστε από διαφορετικά κράτη, από διαφορετικά κόμματα και τελικά εσείς εδώ ε, μας δίνετε όλο το φάσμα μια προοπτική ευρωπαϊκή για τα θέματα που καίνε τους Ευρωπαίους. Οπότε γι' αυτό μας βοηθάτε ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ε, ε μέσω ημών έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και επίσης να πτήσατε την πρακτική αυτών των διερευνητικών ε, αποστολών. Ε, εκεί συναντάτε τους αναφερομένους και ε, επίση έρχεστε σε επαφή με εκπροσώπους των αρχών μέχρι το τοπικό επίπεδο και έτσι ετοιμάζετε τις εκθέσεις σας για όλα αυτά όπως ακριβώς έγινε και για την υπόθεση της Βουλγαρίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το καθημερινό δικό μας έργο Οπότε γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με κάποιες συστάσεις που έχετε διατυπώσει. Έχουμε την πρόσφατη έκθεση του Αντιπρόεδρου Τουργκάη όσον αφορά την εφαρμογή. Είναι εδώ ένα παράδειγμα ε, κλασικό της δουλειά σας. Ε, επίσης, ακόμα και αν αυτό δεν οδήγησε σε μια ε, έκθεση το ότι συνδυάζεται αναφορές για το ίδιο θέμα. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο όσον αφορά τα, αυτά τα αιωλικά πάρκα και τα θέματα που γεννώνται από αυτά. Επίσης, η ισότιμη αντιμετώπιση των ε, αναφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε πάλι να υπάρχουν ε, δίκαιες ε, συνθήκες για όλους όσους ασχολούνται με ένα θέμα. Οπότε είναι σημαντικό το να φροντίζουμε έτσι το περιβάλλον, αλλά υπάρχουν θέματα περίπλοκα και νομικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οπότε το να λαμβάνει κανεί αποφάσει που να είναι σολομόντια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έχουμε όλοι μας την ίδια ε, αυτή πρόκληση. Όπως τα είπαμε και στη διάσκεψη των εμπλεκομένων όλων τον, του, του Ιουνίου. Να δούμε δηλαδή πώ θα εξασφαλίσουμε οι πολίτε να έχουν εμπιστοσύνη στο ότι με το κοινοτικό δίκαιο εμείς εξασφαλίζουμε θετικά αποτελέσματα για αυτούς σε αυτή του ζωή. Βεβαίως, το να κάνετε εσεί καλά τη δουλειά σα, ε, αυτό μα κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι το να προλαμβάνουμε τα προβλήματα για το περιβάλλον όποτε είναι αυτό ε, εφικτό και να μην παρεμβαίνουμε εκ των υστέρων. Οπότε θα πρέπει και εμείς να ωφεληθούμε από την ε, εμπειρογνωμοσύνη που έχετε και εσείς από τη δική μας. Και έτσι μαζί να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τους Ευρωπαίους στο μέλλον. Τώρα, για να έρθω σε κάποια νέα θέματα που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με δύο βασικούς κανόνες όπου μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις. Πρώτα-πρώτα αφορά αυτό το να υπάρχει περισσότερη γνώση των θεμάτων και από την άλλη μεριά ανταπόκριση σε εθνικό επίπεδο. Ε, ενημέρωση, επομένως πληροφόρηση είναι πάρα πολύ βασικό για την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Θα ήθελα επομένως τα κράτη-μέλη να είναι πιο ανοιχτά όσον αφορά την ύπαρξη ε, και το ακριβώς τι γίνεται με τα προβλήματα για το περιβάλλον και για το τι κάνω για να το βελτιώσω. Γιατί αυτό που συνήθως απογοητεύει τους πολίτες είναι το ότι έχουν την αίσθηση ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος ή το κανείς τα κουκουλώνει ε, ή τα, υποβαθμίζει επίτηδες. Οπότε να σας πω ακριβώς τι γίνεται. για ένα θέμα το οποίο το ξέρετε. Ξέρετε όσον αφορά τα τοξικά στο κόρκ της Ιρλανδίας, εκεί στο λιμάνι. Συμφώνησε η Ιρλανδία να γίνει εκεί καθαρισμός και συμφώνησαν ότι ό,τι γίνεται στο μέλλον θα δημοσιεύεται στο Ιντερνετ και έτσι όλοι, όλοι να μπορούν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται και επί Και εγώ ελπίζω τέτοιου είδους προσέγγιση να γίνει ο κανόνας. Και έτσι να μπορούμε να επισημάνουμε το πρόβλημα, να προτείνεται η λύση και να κοινοποιείται τι προσπάθειες καταβάλλονται για να υλοποιηθεί αυτή η λύση. Άρα, όντως θα πρέπει στο ίντερνετ να δημοσιεύει το κάθε κράτος τι κάνει για να υλοποιήσει κάποια οδηγία, να πούμε, όπως η οδηγία για τα ύδατα. Σχετικές εκθέσεις φαίνεται πως βελτιώνεται η κατάσταση για τα ύδατα στην Ευρώπη. Και αυτό για να πίεση των πολιτών αλλά και οικονομικών παραγόντων. Άρα, οι πληροφορίε πρέπει να είναι φιλικέ στο χρήστη και έτσι οι πολίτες να μπορούν να βρουν απαντήσεις γρήγορα στις ερωτήσεις τους. Η ατμόσφαιρα είναι καθαρή. Επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η χωματερή εδώ κοντά. Υπάρχουν επιθεωρητέ. Τι γίνεται, έχουμε περιοχές Natura 2000. Να, τα ερωτήματα. Και επίσης ο βαθμός της ανταπόκρισης είναι σημαντικός. Αυτό σημαίνει το πόσο θέλουν και μπορούν οι αρχές να ανταποκριθούν στα όσα ζητάει ο κόσμος. Πολλέ φορέ τα προβλήματα του περιβάλλοντο έχουν τοπικό χαρακτήρα και πολλέ φορέ γι' αυτό απαιτείται, απαιτείται λύση σε τοπικό επίπεδο. Και εμείς έχουμε, λόγω της φύσης των προβλημάτων, κάποια όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό και θα είναι καλύτερα να γίνεται ό,τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, πώς αυτό μπορεί να το στηρίξουμε. Εγώ έχω κάποιες το κατά νου. Και αυτό οδηγεί σε κάποιες επιθεωρήσεις, ελέγχους, τόσο ώστε να βλέπουμε κατά πόσον έχουμε ε, αξιόπιστη ανταπόκριση επιτόπου. Να λαμβάνουμε επομένως με οργανωμένο τρόπο υπόψη τις καταγγελία των πολιτών και έτσι να βρίσκονται λύσεις ταχύτερα καλύτερη προσβασιμότητα στη δικαιοσύνη γιατί τελικά, τελικά ο δικαστής, ο τοπικός είναι ο πιο αρμόδιος για να παρεμβαίνει σε περίπτωση παρανομίας. Έχουμε την σύμβαση του άρχους και έχουμε τη σχετική οδηγία για την εφαρμογή της. Να, τι μπορεί να μας εμπνεύσει. Όλα αυτά. Ελπίζω ότι θα ζητηθούν στο μέλλον με τους ε, ενδιαφερόμενους και έτσι να φτάσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα έχουμε καλύτερη ανταπόκριση, πώς θα ξέρουμε καλύτερα τα, το, το, τι ισχύει και εδώ τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εκπονηθεί για του χρόνου. Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες χρειάζονται. Και έτσι να βελτιωθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας. Και ελπίζω ότι μπορώ να υπολογίζω στην αμέριστη συμπαράστασή σας. Και είμαι βέβαιος ότι έχετε την εμπειρογνωμοσύνη και αυτό δικαιώνει τη θέση σας και το ρόλο σας. Τώρα να πούμε κάτι συγκεκριμένο για όσον αφορά τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη σχετική οδηγία. Ε, ξέρω ότι όλα αυτά αφορούν ε, την ε, εμπειρία μας και έχουμε πει ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτή η οδηγία δείχνει το πόσο μπορούμε να δουλέψουμε όσον αφορά την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου, αλλά επίσης και έτσι βλέπουμε πώς πιάνουν τόπο οι συστάσεις για το περιβάλλον. Πολλές φορές μιλούμε για κάποια δύνατα σημεία, κάποιες ελλείψεις στα προγράμματα. Και έχουμε τη σχετική οδηγία, EA στα αγγλικά την λέμε, και βοηθάει όσον αφορά μια καλύτερη διαδικασία λήψη αποφάσεων για πολλέ αποφάσεις. Εκεί που έχουμε αντιμαχόμενα συμφέροντα. Προστασία της φύση οικονομική ανάπτυξη. Ε, παντού ισχύουν αυτά. Και σε Βουλγαρία και σε Δανία. Όμως αυτό πολλές φορές δεν μπορεί να ωφελήσει τον κόσμο επιτόπου, όπως πολλές φορές προσδοκούν αυτοί που κάνουν τις αναφορές. Επομένως ακόμα τα πράγματα επιδέχονται βελτίωση, ας πούμε να έχουμε αυτή τη ε, διαδικασία του screening, του, του, ελέγχου των ε, έργων και προγραμμάτων, αυτά τα οποία εδώ πέρα σας απασχολούν και τα έχετε πει και εσείς. Αυτή η συγκεκριμένη οδηγία νομίζω ότι δίνει περισσότερο πεδίο δράση στα κρατημέλη για να μπορούν να δούμε κατά πόσον ε, αυτή η οδηγία μπορεί να συντρέχει για κάποια προγράμματα τα οποία έχουν αποφασιστεί. Πολλέ φορές τα κράτη-μέλη δείχνει εμπειρία. Τα κράτη-μέλη υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες τους, διότι κάποια προγράμματα τα εξαιρώνουν από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η σχετική οδηγία. Και αυτό γίνεται μέσω ακαταλληλών κριτηρίων και οδηγούμεθα έτσι σε κάποιες περιπτώσεις παραβάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, οπότε τα κράτη-μέλη έτσι ε, υπερβαίνοντα καμένα, όμως θα πρέπει από πλευρά μα να κάνουμε ό,τι μπορούμε το ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους ε, παρανομίες. Και είπαμε ότι έτσι θα αναθεωρήσουμε την οδηγία για να προχωρήσουμε σε καλύτερη εφαρμογή της επί τη βάση των μαθημάτων, των συμπερασμάτων που έχουμε αντιλήσει και από τις αναφορές και από ε, τις καταγγελίες και τις αναφορές. Άρα όλα αυτά είναι χρήσιμες πηγές πληροφοριών. Και έτσι φαίνεται το πόσο μπορείτε να βοηθήσετε την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Αφού γκραζόμαστε με τι αγωνίε των πολιτών και έτσι ψάχνουμε τι κατάλληλε λύσει στα πλαίσια τη νομοθεσία και επομένω προχωρούμε σε γυμνά διαβήματα, αναλαμβάνουμε δράση και κατακλείδη. Εγώ θέλω να σα πω ότι η βελτίωση τη ε, εφαρμογή νομοθεσία είναι στην καρδιά αυτού του νέου προγράμματος. Και έτσι προσπαθούμε να δούμε ε, τι θα κάνουμε του, του χρόνου, το δεύτερο εξάμεινο, διότι θα έχουμε την Δανέζικη Προεδρία και την Κυπριακή που θα ακολουθήσει. Και γι' αυτό ελπίζω ότι και εσείς θα βοηθήσετε με δυναμικό τρόπο. Έχετε τις γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά για μας. Θα μας βοηθήσετε και γι' αυτό και εμείς όσο μπορούμε θα συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ κύριε Ποτότσνικ. Δεν είναι μια τυπική ευχαριστία που υποχρεούμε να δώσω αλλά πραγματική, διότι ήταν πολύ, άνοιξε πολλές, ε, πολλά παράθυρα ελπίδα η παρέμβασή σας. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί αυτή η συνεργασία μεταξύ μας. Εσείς απαντήσατε ε, με διάφορα συγκεκριμένα σημεία και προτάσεις για να υλοποιηθεί αυτή η πραγματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και των υπηρεσιών σας. Αυτό μας ικανοποίησαμε μέλη του Κοινοβουλίου αλλά και σαν άμεσους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών. Μας ανακουφίζει, διότι δείχνει μεγάλη ευαισθησία από την πλευρά σας όσον αφορά αυτά που ασχολούν τους πολίτες. Και για να μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ανοίγουμε μέσω τη συζήτηση. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που ζήτησαν να μιλήσουν. Δίνω εν πρώτη το λόγο στο συνάδελφο Μποστινάρου. Κύριε ε, πολύ καλή η παρέμβασή σας, πολύ επίκαιρη. Πριν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις μέσα στα πλαίσια του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεργαστούμε για να μειώσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ αυτών που λέμε στις Βρυξέλλες και αυτών που γίνονται σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσες πολλές αναφορές για περιβαλλοντολογικά θέματα που έρχονται ενώπιόν μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες σημαντικές εκθέσεις σημαντικέ εκθέσει δημοδότηση ή εκθέσει που συζήτηση στην Επιτροπή μας, όπως παραδείγματος η εκθεσει που ζητησα στην επιτροπη μας οπως παραδειγματος η βιοπικιλομορφια για την οποία ήμουν εγώ εισηγητή και μία καλή ακρόση για τη διαχείριση του που οργάνωσε ο αλλά και μια ερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία, στην Βουλγαρία και αλλού. Κύριε Επίτροπε, ένα σημαντικό ερώτημα είναι μπορούμε να βασιστούμε στην ουδετερότητα και αντικειμενικότητα των ε, ερευνών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γιατί αν αυτό γίνεται από τους επενδυτές, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι θα είναι αντικειμενικές και ουδέτερες, ούτως ώστε να εφαρμοστούν τα προϊόντα χωρίς συμπληρωματικό κόστος και χωρίς βλάπη για το περιβάλλον. Στην περίπτωση μεγάλου εύρους έργων θα σύστηνα κύριε Επίτροπε και η αξιολόγηση περιβαλλοντικές ε, ε, των επιπτώσεων και των στρατηγικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων να γίνονται από μια ουδέτερη ε, ε ομάδα. Στη Ρούσια Μοντάνα στη Ρουμανία η ομάδα αυτή εκλήθη ε, ετράφη και λοιπά από τον επενδυτή. Πώς θα είναι ουδέτερη. Δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Μετά, εγώ είμαι συγγητή για το Ταμείο Συνοχής και στο προήμιο της έκθεσης λέγεται ρητά ότι σε ορισμένες συγκεκριμένε περιπτώσεις όπου ο Ριπένον δεν επλήρωσε το κόστος της ρήπανσης, ίσως υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Ταμείο Συνοχής. Θεωρητικά είμαι υπέρ, αλλά στην πράξη κύριε Επίτροπε να είσαστε σίγουρος Κανένα ευρωβουλευτή δεν θα δεχθεί κάτι τέτοιο εάν δεν έχουμε την εγγύηση ότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στρατηγικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα είναι αρκετά ουδέτερες και ισχύς για να αποκλείσουν τις δαπάνε και να μην σπαταλίσουν τα χρήματα του Ταμείου Συνεχής. Είναι σαφές αυτό και μπορώ κάλλιστα να συνεργαστώ με σα πάνω σε αυτό. Τέλο. άλλο ένα ερώτημα. Γιατί η ανακοίνωση που προτείνει ο Επίτροπος Ποτόσνικ στο Natura 2000 τελικά δεν είναι ανακοίνωση του Επιτρόπου αλλά ένα έγγραφο εργασία του των υπολήλων. Γιατί, γιατί δηλαδή αυτό υποβαθμίστηκε κάτι τέτοιο σε ένα επίπεδο που δεν είναι τόσο σημαντικό. Μας είπατε, χρειαζόμαστε εταίρους. Είμαστε στο πλευρό σας ανεφόρων θα έλεγα. Αλλά για να είμαστε στο πλευρό σας είναι ουσιαστικό να μας δώσετε συνεχείς απαντήσεις στους Ευρωπαίους πολίτες, όχι από μια πολιτική ομάδα ή μια άλλη για ένα συγκεκριμένο κράτος και όχι ένα άλλο, αλλά να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα στο Σύλλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πρόθεσή σας για συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο στην αλφας Βάγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχω κάποιες γενικές ερωτήσεις. Εγώ είμαι παρόν για τις δύο αναφορές που αφορούν τη χώρα μου και τα σύνορά μας με την Ιταλία, την περιοχή που βρίσκεται εκεί. Εξέτασα μακροπρόθεσμα τι γίνεται με αυτές τις αναφορές. Ιδίω όσον αφορά <clears throat> τις περιοχές γύρω από τον κόλπο της στεριές της. Έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν προσπαθώντας να απαντήσει στα ερωτήματα που θέσουν ορισμένες οργανώσεις, ιδίω ε, από την κοινωνία των πολιτών, τίθεται η Κομισιόν κάπως σε μια μυθική στάση και είναι σαν να περιμένει να γίνει κάτι κακό για να μπορέσει να κινητοποιήσει το δυναμικό της. Εγώ συμφωνώ με την άποψη που εκφράζεται πλειστάκης από την Εκτελεστική Επιτροπή. Ε, εάν δηλαδή, εάν κάτι αφορά δύο γειτονικέ χώρες, το καλύτερο που θα πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των αρχών των δύο αυτών χωρών. Καμιά φορά όμω, έχουμε την εντύπωση ότι είναι πιο εύκολο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο αυτές χώρες και ε, λιγότερο των τοπικών αρχών και των ε, κυβερνητικών οργανώσεων. Και έτσι οι ομάδες πίεσης, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, είναι τόσο αποτελεσματική η δράση τους που κάποια φορά έχει κανένα την εντύπωση ότι η διοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αντιταχθεί. The Commission have the instruments to play, uh, Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι τα μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Κομισιόν για να παίξει ένα πιο αποτελεσματικό, ενεργό, ισχυρό ρόλο στις περιπτώσεις αυτές. Και οι πολίτες που ζητάνε από την Επιτροπή να παρέμβει, τι περιμένουν από την Επιτροπή. Υπάρχει κανένα σχέδιο να βελτιωθεί η δυνατότητα ανταπόκρισης της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Βιλό. Ausführungen. Ich möchte nicht von meinem Land sprechen. Εγώ δεν θα μιλήσω για τη δική μου χώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα φιλικά σας λόγια και ότι είμαστε εταίροι, αλλά θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν είμαστε μόνο ε, σύντροφοι και εταίροι, αλλά είμαστε και εκείνοι που καταδεικνύουν αυτά που δεν ε, πάνε σωστά για όλα τα στραβά, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα εκεί που δεν υπάρχει η σωστή νομοθεσία. Η περιβαλλοντική πολιτική εδώ έχει διάφορους ρόλους. <clears throat> Καταρχήν πολλές φορές α, επαναλαμβάνεται η συζήτηση που γίνεται στις διάφορες χώρες χωρίς εδώ να βλέπουμε ότι η Κομισιόν η Ευρώπη να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα. Άλλες φορές το περιβάλλον χρησιμοποιείται σαν είσοδος, δημόσια την υπόθεση της, του αγωγού μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, όπου υπήρχαν προβλήματα στον αφορά τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσει και που η έρευνα αυτή κατέληξε εδώ στη χέρια μας. Ή παραδείγματος χάρη το, ε, η νομοθεσία προστασίας ε, των ακτών της Ισπανίας όπου εισάγονται πρότυπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα αυτή. Μετά έχουμε τις υποθέσεις όπου το περιβάλλον είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι ελλείψεις που παρουσιάζονται δεν καταδεικνύουν ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Έχω και κάτι το συγκεκριμένο να σας πω, όπου θέλω να μου απαντήσετε είπατε ότι η ενιαία νομοθετική δέσμευση είναι το κλειδί για μια ομοιόμορφη εξέλιξη, Λένε και το κλειδί και για τον πολίτη. Γιατί αν ο πολίτη βλέπει ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο από μια περιοχή στην άλλη και από ένα κράτο στο άλλο, χάνει αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ διαβλέπω κάποια προβλήματα όταν ε, εργάζεται με συστάσεις όπως θέλετε γιατί έχουμε εδώ μια διαφορά μεταξύ ε, Κομισιόν και ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διάφορες αυτές νομοθετικές πράξεις οι οποίες δεν είναι και πολύ δεσμευτικές όπως οι συστάσεις η κατεξιοντότηση πράξης είναι κάτι που δεν ικανοποιεί πάρα πολύ το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη μορφή λέω πάντα Λοιπόν, γρήγορη νομοθεσία είναι καλή και η αργή είναι κακή. Το ίδιο είναι και με τις αναφορές. Η γρήγορη αναφορά είναι καλή, η αργή είναι κακή. Το θέμα είναι πώς νομοθετούμε, πόσο γρήγορα νομοθετούμε και κατά πόσο νομοθεσία πάνε από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω τα εξή τέσσερα. Καταρχήν, έχουμε στις αναφορές ένα χρονικό χάσμα. Θα ήθελα να προσπαθήσετε να συντονίσετε το, το δικό σας, ε, τους δικούς σας ε, συνεργάτες με εμάς για την πρόσθεση των αναφορών. Δεύτερον, θα ήθελα να με βοηθήσετε μέσω του Συμβουλίου, ούτω ώστε οι χώρες ε, μέλη να συνεργάζονται καλύτερα μαζί μα. Ορισμένοι το κάνουν ήδη εδώ όταν συζητείται κάποια συγκεκριμένη ανάφορα, άλλοι σε εξαφανίζονται. Θα ήθελα να είναι καλύτερη η αντιμετώπιση αυτού του θέματο, τη ε, παρουσία των κρατών μελών. Τρίτον, δεν έχω πάντα την εντύπωση ότι υπάρχει συμμεταχείριση των κρατών μελών. Έχω την εντύπωση όταν τοποθετούνται εδώ ε, οι υπάλληλοι τη Κομισιόν, εάν ο εχθρό είναι μεγάλο και ωραία η κυβέρνηση, δεν θέλουν να εφαρμοστούν. Αν όμως η χώρα είναι μικρή και κακή η κυβέρνηση, όλοι είναι πολύ τολμηροί. Και εκεί περιμένουν να υπάρχει πιο ομοιογενής και ενιαία αντιμετώπιση. Και τέταρτον, η νομοθεσία εκ των κάτω προς τα πάνω. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα πάντα εκ των άνω προς τα κάτω σε όλες τις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι νόμοι να σηκώνουν από κάτω προς τα πάνω και γι' αυτό θα ήθελα η Κομισιό να κάνει μια μελέτη πώς η Προσφυγέ στο Λουξεμβούργο για προκαταρκτικές αποφάσει ε, μπορούν να τύχουν επεξεργασίες στα κράτη-μέλη. Έχω την εντύπωση ότι πολλέ, πολλά δικαστήρια λένε δεν χρειάζομαστε το Λουξεμβούργο, μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας και αυτό είναι πάρα πολύ ε, χρονοβόρο και κοστίζει και ακριβά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Ριβελίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και επίτροπε. ευχαριστώ. Είμαι ένα πολίτης από την Νάπολη. Γεννήθηκα στην Νάπολη, είμαι Ευρωπαίο, είμαι κοινοβουλευτικό ε, Ευρωβουλευτή και ο Επίτροπός μου ε, ε, είσαστε επίτροπό μου, επίτροπο για το περιβάλλον και ζητώ για μια άπαξη απαντό να λύσετε το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων ε, στην Νάπολη. Οι πολιτικοί φορεί ντόπιοι ήταν ανίκανοι να το λύσουν και η Ευρώπη όμω που παρενέβη συχνά ε, με μεθόδους πολύ ασαφείς και με ελάχιστα αποτελέσματα. Θα ήθελα να επαναλάβω κάποια θέματα σημαντικά. Το πρώτο απ' όλα θα πρέπει να εξηγενθεί η περιοχή, θα πρέπει να χρηματοδοτήσει η Ευρώπη το να καθαριστεί η περιοχή. Είναι κάτι που οφείλεται και σε απαταιώνες Ευρωπαίους και Ιταλούς ε, που εκμεταλλεύτηκαν το έδαφος μας. Γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα. Δεύτερον, χρειάζεται παρέμβαση ώστε να γίνει σεβαστή το σχέδιο για τα απόβλητα που η περιοχή της Καμπανίας παρουσίασε και απεδέχτη η Ευρώπη. Ένα σχέδιο λοιπόν για τα απόβλητα που προβλέπει ένα ολοκληρωμένο κύκλο για τα απόβλητα, μια συλλογή διαφοροποιημένη των αποβλήτων και την κατασκευή ενό κλειβάνου τελευταίας γενιάς στην πόλη. Ο νέος δήμαρχος της ε, Νάπολη, ο Δεματζίστρης, που ε, πριν από 6-7 μήνες δήλωσε ότι σε 3 μήνες θα είχε οδηγήσει τη διαφοροποιημένη περισυλλογή στο 70% των αποβλήτων, κάτι που ποτέ δεν συνέβη σε καμία πόλη του κόσμου, σήμερα ε, έχει χρεοκοπήσει αυτή η προσπάθεια, διότι έχω τα επίσημα στοιχεία που σας έδωσα, που, που βγαίνουν και στις σημερίες εφημερίδες της περιοχής, που δείχνουν τα στοιχεία ότι την τελευταία περίοδο, την πρόσφατη περίοδο, η συλλογή διαφοροποιημένη των αποβλήτων στην περιοχή του, της Νάπολης μειώθηκε από το 2009 μέχρι το 2011 κατά 2%. Αλλά συνάδελφοι της Επιτροπής Αναφορών, που όπως εγώ εδώ και ένα χρόνο συμμετείχαν σε, επιστολή, σε αποστολή στην Καμπανία, θα θυμούνται ότι στην Ομαρχία ε, παρουσιάστηκαν επίσημα στοιχεία όσον αφορά τη διαφοροποιημένη ε, συλλογή αποβλήτων στην Άπολη που ήταν σε ποσοστό περίπου 22%. Σήμερα έχουμε στοιχεία πολύ κατώτερα, πολύ κατώτερα αποτελέσματα παρόλο που ο Δήμαρχος Δεματζίστρης όλο λέει λόγια, λόγια, ανοησίες και ανόητα στοιχεία. Ο ίδιος Δήμαρχος και σας παρουσίασε σχετική τεκμηρίωση και όλα είναι σαφή στην τεκμηρίωση δεν θέλει, δεν επιθυμεί να υπάρξει ε, θερμοκλίβανο στην Νάπολη και φρόντισε ο, τελικά να μην υπάρξει υποψήφιο στο διαγωνισμό. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει ολοκληρωμένος κύκλος για τα απόβλητα και συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή ενός ε, κλιβάνου για τα απόβλητα. Τέταρτον, ο Δήμαρχος σήμερα θέλει να εξαγάγει στην Ολλανδία τα απόβλητα. Κάτι που ήδη επεκρίθη από την Ευρώπη όταν ο προηγούμενος επίτροπος ο Μπασολίνη είχε εξάγει τα αποβλήτα στη Γερμανία και αυτή η εξαγωγή των αποβλήτων που εδώ στο Κοινοβούλιο βρίσκει μεγάλη αντίθεση και παρουσιάστηκε και ερώτημα του Ολλανδού συναδέλφου Ντεάν σχετικά με το θέμα, είναι κάτι που αντιβαίνει αυτή η πρόταση, αντιβαίνει τι ευρωπαϊκέ οδηγίε. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε, ζητώ από εσά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν στην πόλη της Νάπολης ούτω ώστε να καταλάβει σε ποιο βαθμό, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατάσταση και πόσο επίγονη το θέμα των αποβλήτων. Είναι μια, πρόβλημα μιας πόλης, της Νάπολη, μιας ευρωπαϊκής πόλης που είναι και δική σας πόλη ε, και θα πρέπει να προσπαθήσετε να τη βοηθήσετε διότι οι Ναπολιτάνοι είναι και συμπολίτε Δεύτερον, εσείς Επίτροπε θα πρέπει να εξακριβώσετε κατά πόσο υλοποιείτε το σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Ιταλία και έγινε αποδεκτό από εσά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτό το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε, εάν ο Δήμαρχος Δεμαντζίστρης δεν σέβεται αυτό το σχέδιο, εάν η διαφοροποιημένη περισυλλογή των αποβλήτων δεν ξεκινήσει, θα πρέπει να παρέμβετε έναντι της Ιταλικής κυβερνήσεως, ώστε να υπάρξει Ιταλική νομοθεσία που θα πρέπει ε, να εφαρμοστεί ούτω ώστε η κοινότητα της Νάπολης ε, θα πρέπει να, να κινηθεί και να απομακρύνει το Δήμαρχο από τη θέση του. Εάν δεν μπορέσετε να το κάνετε αυτό, εγώ σαν Ευρωβουλευτής θα πρέπει να ζητήσω από τον Υπουργό μου του Περιβάλλοντος, εσείς κύριε Επίτροπε, οι διευθύνσεις σας να, παρουσ, να παρουσιαστεί εναντίον σας μία ε, πρόταση μορφής Διότι εσείς είστε ο Επιτροπός μου, εσείς είστε ο υπουργό μου, εσείς είστε εκείνος που θα πρέπει να εφαρμόσει τα σχέδια ε, τα οποία έχουν υποβληθεί και από εσά θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ συνάδελφα να υπενθυμίσω ότι στις 10.30 πρέπει να μας εγκαταλείψει ο Επίτροπος και για να του δώσουμε δυνατότητα σα απαντήσει θα πρέπει να είμαστε πιο συνοπτικοί. Ο κύριος Γιάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Äh, Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Επιτρόπος με τον οποίο είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος. Δεν νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό το να ε, έχουμε αυτές τις αναφορές για τις περιπτώσεις της ε, καταπατητήσεως δικαιωμάτων. Θέλουμε επομένως εμείς εδώ να μπορούμε να ε, κρίνουμε με τρόπο αμερόληπτο, να προσπαθούμε βέβαια να βοηθήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα το πράσινο και το κόκκινο. Πράσινο σημαίνει ότι δεν παραβιάζει την νομοθεσία. Κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε κατάφορες παραβιάσεις αυτής. Οπότε θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται μετά κρατη Τι κάνουν τα Για να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτέ τι αναφορέ που έχουν το χρώμα το κόκκινο, <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, διαπιστώνουμε παραβιάσεις τη νομοθεσία. Οι αναφερόμενοι έρχονται και μας λένε εντάξει διαπιστώνετε την παρανομία και τι κάνετε παρακάτω. Δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση και να ενεργούμε ταχύως όποτε έχουμε σημαντικές παραβιάσεις του δικαίου. Έχουμε για τι το χρώμα το κίτρινο. Εκεί όπου είναι αβέβαιο το τι συντρέχει. Εκεί έχουμε οριακές περιπτώσεις. σχέση με την νομοθεσία. Πολλές φορές προτείνουμε τροποποίηση της νομοθεσίας. Το πρόβλημα όμως με αυτές τις κίτρινες αναφορές είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης των πραγμάτων. Να μπορούμε να ξέρουμε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τα όσα γίνονται, να διαπιστώνεται το τι κάνουν τα κρατημέλη. Όμως, μετά από το σχεδιασμό του επομένου διαβήματος, έχουμε χρήματα και θέσεις απασχόλησης που διακυβεύονται. Άρα πρέπει κανείς να παρακολουθεί το τι γίνεται. Έχει δίκιο, κύριος Βίλαντ τα κρατημέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται και να ακούει τη φωνή τους εδώ ή στην Επιτροπή των Αναφορών. Ευχαριστώ, λέει κυρία Όκεν. Χαίρομαι που και οι πράσινοι έχουν επίσης το λόγο. Πολύ καλά. εξεπλάγει Ακόμα και οι γυναίκες περιμένουν στη σειρά, αλλά εδώ δεν υπήρξε πρόβλημα. Ευχαριστώ, Επίτροπε τότε για την παρουσία σας. Είναι σημαντικό που φαίνεται ότι γνωρίζετε πόσο συμμετοχή των πολιτών είναι σημαντική. Εδώ εμείς εκπροσωπούμε πρώτα απ' όλα τους αναφέρονται στους πολίτες. Θα επικεντρωθώ επί της ε, συμβάσεως του όρχους, της παλαιάς. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες να εφαρμοστεί το τρίτο τμήμα όπως και τα δύο πρώτα χρειάζεται για να βελτιωθεί η κατάσταση για τους πολίτες. Για να και συμμορφωθούν και αυτοί, να μας δίνουν σωστές πληροφορίες. Χωρίς τους πολίτες δεν μπορούμε να κινηθούμε. Το ξέρετε κι εσείς ότι γίνεται πολύ σημαντική δουλειά για να εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. πολύ συχνά το αποτέλεσμα που μας παραδίδεται είναι έξοχο. Και το θέμα της διαφάνειας είναι σημαντικό. Οι διαδικασίες κατά παράβαση πρέπει να είναι διαφανείς και το ταχύτερο δυνατόν. Μιλάμε για την ασφάλεια και την πιστοσύνη των πολιτών που πρέπει να φροντίσουμε. πρέπει να το φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας λείπει η διαφάνεια. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στοιχεία. Γίνεται μάχη για το κανονισμό 1049. Θέλουμε υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να γίνει ιδέως αναβάθμιση σύμφωνα τη νέα νομοθεσία και τη συνθήκη και τη σύμβαση και την παλιά. Ελπίζω ότι η συνάδελφος Εντρίν θα μιλήσει και εκείνη για τη Natura 2000. Και το δεύτερο σημείο αφορά τα απόβλητα. Συνεχώς το βρίσκουμε μπροστά μας το θέμα. Οι χρήσιμες εναλλακτικέ πέρα από την καύση εξετάζονται. Και είναι τα πάντα στη χώρα μου. Είναι πολύ καλοί καυστήρες η κλίβανη. Είχαμε και την έκθεση του Γάι που εκεί είδαμε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα, να μην καίγονται απλώς. Υπάρχουν κομψότατες τεχνολογίες και σχέδια, ούτως ώστε και απόβλητα να τα επεξεργαζόμαστε με πολύ φθηνό τρόπο να παίρνουμε αέριο, να χρησιμοποιούμε σαν καύσιμα αυτά τα απόβλητα. Μετά μπορώ να σας μιλήσω εκτενέστερα, αν θέλετε να μάθετε. Και ο αρμόδιος φορέας μας δώσει τις πληροφορίες. Αντί να χρησιμοποιούμε την ευρύτατα διαδεδομένη καύση που καίμε τα πάντα, να κάνουμε άλλη χρήση, γιατί καίμε και πολύ σημαντικές ύλες, όπως φόσφορο. όπως και στην Άπολη. Θέλουμε συμμετοχή των πολιτών. Χωρίς συμμετοχή τους δεν θα πετύχουμε. Δεν θα βρούμε βιώσιμη λύση όσον αφορά τα απόβλητα. Και στην Άπολη και αλλού είδαμε ότι όταν δεν συνεργάζονται ε, πνίγονται τα σκουπίδια τελικά. Και είναι ένα πρόβλημα που όλο και περισσότερο το βρίσκουν μπροστά μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Μπελέτ, δύσκολο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτρο, θα είναι δύσκολο να απαντήσεις όλες αυτές τις ερωτήσεις σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Εκτός αν έχετε περισσότερο χρόνο εδώ. Εγώ φαντάζομαι να θα δώσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την Natura 2000. Θα μιλήσω πολύ σύντομα. 20-30 χρόνια που δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την ποικιλομορφία. Και βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση των κρατών μελών. <coughs> Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα αυτή τη εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη, <coughs> ούτω ώστε επιτέλου αυτά να εκπληρώνουν τι υποχρεώσει του για την Natura 2000 και την ποικιλομορφία. Σήμερα όμως θεωρώ ότι όλα τα μέσα στη διάθεσή μας και στη διάθεση της Κομισιόν δεν χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιβεβαιωθεί η πολιτική βούληση του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο είναι ε, το χρηματοπιστωτικό. Ε, μέσα στις απλή στρατηγική 2020 είχε αναφερθεί ότι θα υπάρχει μια μελλοντική ανακοίνωση της Κομισιόν για την χρηματοδότηση για το Natura 2000 και το, την ποικιλομορφία. Για φέτος είχε προαγγελθεί αυτή. Πότε θα μας την παρουσιάσετε, τι γίνεται όσον αφορά επίσης για τη διατηρησία, για τις πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν σήμερα ενώπιον της ε, ε, Επιτροπής Αναφορών για καταπάτηση του κοινοτικού δικαίου είναι σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης για την ποικιλομορφία και Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την καταστροφή της ποικιλομορφίας αυτής. Και τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία, αναρωτιέμαι ποια είναι η λίστα ανάλυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά Εναλλακτικέ προτάσει των κρατών μελόφθων, ίσω το σημείο το πιο δύνατο των προτάσεων που έχουμε μπροστά μας. Τι προτείνει η Κομισιόν για να προωθήσει τα κράτη-μέλη να μας παρουσιάσουν εναλλακτικά μέσα. Και έχω και μια άλλη ανησυχία στα πληθές ε, Αν ρωτιέμαι τι γίνεται όσον αφορά αφενός ε, την καταπολέμηση των ε, κλιματολογικών αλλαγών και την καταπολέμηση της απόλυτης βιοποικιλομορφίας. Πού βρίσκεται η διατησία μεταξύ των δύο και δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή ο στόχος της καταπολέμησης της αλληλεγγύης του κλίματος να θεωρηθεί πιο σημαντικός από την διατήρηση της ε, βιοποικιλομορφίας. Δεν θα ανατήσω λοιπόν ποιο ε, κάνει τη διατησία αυτή και ποια είναι η σχέση την ισχύω. Ευχαριστώ κύριε Μέρκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω πέντε θέματα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Είχαμε ήδη την ικανοποίηση να αλλάξουμε συχνά απόψεις. Δεν θα επαναλάβω αυτούς very important to have a format on how to deal with ε, θα ήθελα ε, να μου πείτε κάτι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα των αποβλήτων. Γιατί πήραμε τόσες πολλές αναφορές, ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα, όπως αναφέρεται στην έκθεση του συναδέλφου Ιντογκάη είναι πολύ καλό νομίζω να έχουμε ε, μια μορφή αντιμετώπισης κάθε χώρας, κάθε περιοχής ε, όταν προσιάζεται το πρόβλημα αυτό. Επίσης, είναι δίκαιο αυτές οι περιοχές ή οι χώρες να έρχονται ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών για αυτή, αυτό. Είναι ένα θέμα που αφορά πολύ τους ε, πολίτες και όταν εμείς υποδεχόμαστε τους αναφέροντες. Δεν θέλουμε να κάνουμε δίκη εδώ, αλλά να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Θα ήταν καλό λοιπόν να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό σε αναφορών. Τρίτον, θεωρώ ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να βρεθεί μία μέθοδος για να υποστηριχθούν οι περιφέρειες όταν κινούνται προς περισσότερη αηφορία και καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής για, τις, ε, για τα απόβλητα. Γιατί πολλές φορές οι περιφέρειες δεν ξέρουν τι να κάνουν, πόσο προσωπικό θέλουν, τι προσωπικό θέλουν, τι εκπαίδευση πρέπει να έχει αυτό για να μπορούν να εφαρμόζονται οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι εποπτεία δηλαδή μόνο, αλλά και βοήθεια. Τέσσερα. Χρειαζόσαστε νομίζω μια στρατηγική παρέμβαση. Ε, έχετε βέβαια, το ξέρουμε, αλλά ποια είναι τα βήματα που αναλαμβάνετε, σε ποιες περιπτώσεις. Πότε δηλαδή έρχεστε σε επαφή με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χάν, για πάγωμα των περιφερειακών ταμείων. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται κάθε φορά και Τέλος, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναείπα στο παρελθόν πολλές φορές, η Επιτροπή μας έχει συζητήσει το θέμα των χωματορών. Ξέρω ότι θα μου πείτε, όλες οι περιφέρειες της Κομισιόν δεν πρέπει να ε, τύχουν απαγόρευσης των χωματορών. Αλλά εντάξει, κλείνουμε μερικέ πόρτε, πρέπει να ανοίξουμε άλλε. Εάν δεν έχουμε όμως απαγόρευση δεν θα φτάσει η Ευρώπη εκεί που θέλουμε, δηλαδή σε ένα πιο βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο Ποτότσνικ, ούτω ώστε να δώσει απαντήσεις και ελπίζω να τα καταφέρει να τα κάνει στα λίγα λεπτά που τα απομένουν. Ίσως μετά θα ακολουθήσουν γραπτές απαντήσεις αν θέλει κάτι τέτοιο ο κύριος Επίτροπος lot of Πολλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνοπτικός γίνεται. Αν αφήσω κάτι εκτός ή λησμονήσω κάποιον από εσάς ή κάποια ερώτηση, σας παρακαλώ. Έχω συναδέλφους εδώ στην αίθουσα που θα απαντήσουν όπως είπατε. Να ξεκινήσω προσπαθώντας να εξηγήσω με ποιο, το, ποιο τρόπο προσπαθούμε να κινηθούμε όταν αντιμετωπίσουμε τα κράτη-μέλη. Όλη η ιδέα βεβαίως όσων συζητούμε, αναφορές, παραβιάσεις και λοιπά, νομοθεσία, όλα αυτά έχουν σαν σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος επιτόπου. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα και ό,τι κάνουμε το εξετάζουμε από αυτή την ε, οπτική γωνία. Όταν ασχολούμεθα λοιπόν με τα κράτη-μέλη, ακολουθώ ένα σύνθημα, προσπαθώ να το ακολουθήσω. Να, να είμαι επικοδομητικά αυστηρός και μαστηρότητα επικοδομητικό. Λοιπόν, προσπαθώ να παίξω το ρόλο του θεματοφύλακα των συνθήκων. Αυτή είναι η υποχρεωσή μου. Και πολλές φορές οι υπάλληλοι με τους οποίους συζητώ δεν είναι ικανοποιημένοι και πολλές φορές έχω κάποιες δυσάρεστες συναντήσεις όταν συζητούμε αυτά τα θέματα, αλλά αυτό είναι ο ρόλος μου και σας εγγυώμαι ότι θα δραματίσω αυτό το ρόλο, θα παίξω αυτό το ρόλο μέχρι τέλους. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ ό,τι καλύτερο για να έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών μελών. Είτε είναι μεγάλα είτε μικρά κράτη-μέλη. Στο επίπεδό μου σας εγγυώμαι ότι επειδή προέρχομαι από μικρή χώρα προβληματίζομαι όλος ιδιαίτερα αυτό το θέμα και δεν θα αντιμετωπιστεί κάποιος διαφορετικά όσο εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το τομέα. Καμιά φορά ίσως δημιουργείται εντύπωση ότι αυτό δεν αληθεύει, αλλά τίποτα δεν γίνεται εκ προθέσεως ή σκόπιμα όταν συμβαίνει αυτό το πρόβλημα. Αντιθέτως, πολλές φορές όταν κάποιος θέλει να κινηθούμε ταχύτερα ή με διαφορετικό τρόπο, πρέπει να φροντίσουμε ότι ακολουθούμε μια οριζόντια προσέγγιση. Οι σχέσεις με τα κράτη-μέλη όταν ασχολούμαστε με τα θέματα των κρατών μελών, το σημαντικότερο είναι, και δεν έχω και επιλογή άλλωστε, είναι λοιπόν να αναπτύξουμε σχέση εμπιστοσύνης. Αν κάτι το οποίο μου αναφέρεται από υπαλλήλους, από εκπροσώπους ή ασδήποτε κυβερνήσεως αμφισβη... λέγεται, αμφισβητείτε, συζητείτε. Και αν λαμβάνουμε μια καταγγελία, εμεί ξαναρωτάμε, θέτουμε το ερώτημα. επιστρέφουμε και λέμε στα κρατη έχουμε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε αυτό και επί τη βάση αυτού προσπαθούμε να κρίνουμε με δικαιοσύνη. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά την εμπιστοσύνη. Εκεί πρέπει να βασίσουμε τη σχέση μας. Είμαστε εταίροι. και είστε μέσω ανακοινώσεως ή οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το κοινοτικό δίκαιο το προσπαθούμε μέσω συμφωνιών συνεργασίας με κάθε κράτος μέλος να το κάνουμε αυτό, όπου εντοπίζουμε από κοινού τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν και μαζί προσπαθούμε να βρούμε σωστές λύσεις. Η ιδέα είναι να αλλάξει πραγματικότητα επιτόπου, διότι αν δεν γίνει αυτό, αν προσπαθήσουμε να ε, δείξουμε τη δύναμή μας ε, εδώ και εκεί, δεν θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα, την εξουσία, τη δύναμη σε όλους τους εμπλεκομένους σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα να κάνουν αυτό που πρέπει. Σε εθνικό επίπεδο καταβάλλονται προσπάθειες στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα προβλήματα σε κεντρικό επίπεδο και το ξέρετε πολύ καλά. Διότι τις πληροφορίες μας δίνετε κι εσείς. Αυτό το αναφέρατε. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν το θέμα για την, για την ε, ανακοίνωση, κοινοποίηση και τη χρηματοδότηση του Natura. Θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση του Natura και στο ιστορικό. Η επιτυχία του Natura εξαρτάται από δύο κρίσιμα θέματα. Την καλή διαχείριση και τη σοβαρότητα της χρηματοδότησης. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. πιθανότατα δεν παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις, αλλά προσπαθήσαμε πάνω να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά τη διαμόρφωση προτάσεως για την κοινή ερωτική πολιτική και για να είμαι σύντομο. Τα χρήματα που προέρχονται από την ΚΑΠ σε τρέχουσες τιμές είναι 20 δις στην παρούσα δημοσιονομική προοπτική και στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική πάνω από 100 δις. δεν θα πληρώνεται ο Γιώργος αν η δραστηριότητά του δεν θα συνδέεται με πράσινες δραστηριότητες. Είναι σημαντικότατο αυτό, υψίστης της σημασίας, διότι οι γεωργοί είναι εκείνοι που διαχειρίζονται τη γη και τα δάση για μας. Έχουν στα χέρια τους τα τρία τέταρτα των γεών των εδαφών στην Ευρώπη. Και έχουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη βιοπικιλότητα με την ε, ποιότητα των υδάτων ε, με το έδαφος, με τη γη. Οπότε όλα, αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε να λυθούν και γι' αυτό το λόγο και εμείς προωθούμε τόσο έντονα αυτή την έννοια του, του, του, του κοινού, του δημοσίου αγαθού. Οπότε πάνω σε αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και εκτός από αυτού του είδους την, την άμεση ενίσχυση, τους δίνουμε ενίσχυση για αυτό το κοινό καλό. Και να η πρότασή μας και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να έχουμε δυσκολία βέβαια αυτό να περάσει τόσο στο κοινοβούλιο όσο, τόσο και στα κρατημέλη πάλι νομίζω ότι είναι σημαντικό όμως να το δούμε γιατί πρόκειται για ένα νέο βήμα, νέα φιλοσοφία όσον αφορά το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα όλα αυτά που συζητούμε επίσης. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει να κάνει και με την πολιτική της συνοχής την πολιτική αλίας. Δεν ξέρω. Η κυρία Δαμανάκη νομίζω ότι είναι κάποιος ο οποίος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά την έννοια ε, της ε, βιωσιμότητας και της αηφορίας και νομίζω ότι το έργο της είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε επομένως όλα αυτά τα τα, τα θέματα, όλα αυτά τα στοιχεία, ούτως ώστε θα πρέπει να τα συνδυάσουμε για να δούμε τις δυνατότητες ε, χρηματοδότησης. Πολλές φορές πρόκειται για άμεση εκταμίευση, αλλά πολλές φορές κρίνεται αυτό από την περιφέρεια ή από τα κράτη-μέλη και έτσι. Ε, βλέπουμε κατά πόσο πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα και να, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, οπότε έχουμε αυτή την ανακοίνωση και έχουμε αυτή την ε, κατάσταση. Δεν ξέρω θα είναι τι τελικά προεκτώσει. Όμω αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να συγκεράσουμε όλα τα στοιχεία και έτσι τελικά να μπορεί κανεί να καταλάβει σαφώ πώ, πού προσφέρονται ευκαιρίε, πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Αλλά ανοίξαμε όλε αυτέ τι πόρτε οι οποίε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή στο μέλλον για να εκμεταλλευτούμε όλε αυτέ τι ευκαιρίε. Παρακάτω. Έχουμε κάτι το οποίο το έθιξε ο Ιβο Βάγκελ. Ναι, ορθώς είπατε ότι έχουμε κάποια διλήμματα σε σχέση με το τι γίνεται για τη διάρκεια της Εάν ρίξετε μία ματιά σε αυτή την ε, ιστορική εξέλιξη της ε, περιοδικής αξιολόγησης πριν έχουμε κάποιο είδους ε, απόφαση, δεν γινόταν πριν την απόφαση αξιολόγηση. Επομένως, Και μόνο που υπάρχουν, ε, υπάρχει αυτό σαν, σαν, θεσμός είναι να βήμα προ τα μπρο. Όλα αυτά θα πρέπει να ισχύσουν και όπω ξέρετε φαίνεται και από τη δική σα δουλειά ότι δεν συμφωνούν με τα κράτη-μέλη. Πολλέ φορέ καταχρώνται του ρόλου τους, των δυνατοτήτων τους και δεν ε, κάνουν αυτό που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Και επομένως Το θέμα της διαφάνειας τι σημαίνει. Ότι όλα τα οποία γίνονται σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρει κανείς αν γίνεται αυτά τα πράγματα ή όχι. Να, τι γίνεται όσον αφορά την ε, αντικειμενικότητα την αμεροληψία, τη διαφάνεια. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε κατά πόσον κάποιο θέλει στα σοβαρά να δει μια πρόταση, μπορεί να κρίνει. Γιατί πρόκειται για μια πρόκληση, είναι μια δυνατότητα που προσφέρεται. Ξέρω επομένω πώς έχει η κατάσταση. Ξέρω ότι τα πράγματα δεν είναι ιδιώδη και για αυτό και εμείς συνεχώς Πρώτα να δούμε πώς η οδηγία αυτή που EA θα γίνει πιο αποτελεσματική και όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για το περιβάλλον, για τον κόσμο. Τώρα, μία-μία φράση μόνο. Όχι. Δεν θέλω να μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες και εξατομικές για περιπτώσεις. Σχέση με αυτούς τους τερματικούς σταθμούς στην Τεργέστη. Ανέκαθεν προσπαθούμε να είμαστε δυναμικός, ενεργός παράγων, παίκτης. Ίσως περισσότερο από τον μέσο εμπλεκόμενο. Ξέρετε, ακόμα και στη δική μου χώρα μας προσέχουν πάρα πολύ. συνεχής ροή πληροφοριών και ενημέρωση από όλου. Και έτσι βλέπουμε κατά πόσο υπάρχει η σωστή εξολόγηση των πληροφοριών. Βλέπουμε τι γίνεται με τι πληροφορίες, γιατί επίσης για την διαμόρφωση ενένεσης αυτή η οδηγία λέει ότι κατά την διαβούλευση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις. Και όταν κάποιο δεν κάνει αυτό το οποίο δεσμεύτηκε να κάνει, θα πρέπει να και το εξηγεί. Δεν είμαστε όμω σε αυτή τη φάση. Ανέκαθεν, έχουμε όλο τον κόσμο ενθαρρύνει. Αυτή η διαβούλευση, επομένως που έγινε, προβλεπόταν από την ε, οδηγία Το ίδιο έχει και για την ανακοίνωση, στην οποία προέβημε. Σας εγγυώμαι ότι παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις. Και η εξωτερική μας κρίση διαμορφώνεται πάντοτε με βάση αυτά τα δεδομένα. Push also in when we discuss that issue. Όταν τα συζητάμε πάντοτε. Έχω υπόψη ότι δεν πρόκειται μόνο για του συγκεκριμένου τερματικού σταθμού. Εγώ κάθε φορά λαμβάνω υπόψη ότι το περιβάλλον τελεί υποπίεση. Εκεί, στην Βόρεια Αδριατική. Για μένα, επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σοβαρή συνεργασία των κρατών που βρέχονται από την Βόρεια Αδριατική. Να καταλάβουμε ότι πρόκειται για στρατηγική σημασία θέμα το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει, να σημαδεύει ό,τι κάνουν στο μέλλον. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία Ανδριατικής ε, Ιωνίου να έρθει και να συντεριάξει με την στρατηγική για τη Βαλτική, για τη Βόρεια Θάλασσα κλπ. Γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα θέματα να, να, να ρυθμιστούν αλλιώ. Να τα κάνει κανεί από τι Βρυξέλλε, όχι. Θα πρέπει κανεί να μπορεί να κάτσει το τραπέζι με αυτούς που τους αφορά το θέμα άμεσα, να του δώσει να καταλάβει πόσο θέμα σημαντικό, πόσο ευάλωτο είναι τελικά το περιβάλλον. Harmonization, um, Mr. Villand, uh, unfortunately has to leave, but uh, he has good excuse. Ένα uh, άλλο θέμα. Νομίζω το θέμα αυτό το οποίο είπατε και το πώς θα διεκπαιρεώσουμε ταχύτερα είναι σοβαρό για να είμαι ειλικρινής μαζί σας και εμείς προβληματιζόμαστε για το πώς θα επιταχύνουμε τη διαδικασία. Από την άλλη μεριά, βέβαια, επίσης, θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τη διαδικασία της παράβασης τα καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Γι' αυτό πριν που, τότε που εργαζόμουν με, για επιστημονικά θέματα και θέματα έρευνα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πραγματικά ό,τι μπορούμε. Χρησιμοποιούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Έχουμε τώρα 470 σε σχέση με, την, με όσους ασχολούνται με το κλίμα με την γραμματολογική μεταβολή δηλαδή. Και έχουμε τώρα καινούργιες προκλήσεις συνέχεια. Καινούργιες προκλήσεις και όλα θα αντιμετωπιστούν στην ώρα τους. Πάντως, ε, όντως, η συγκυρία είναι δύσκολη. Και αν έχετε κάποιες ε, ιδέες στρατηγικού χαρακτήρα για το πώς θα βελτιωθεί η συνεργασία μας, θα έτοιμοι να τις ακούσουμε. Δεν υπάρχουν όμως εύκολες λύσεις. Ποιο κ. Βίλαντ επίσης μας είπε ότι δεν θα πρέπει μόνο από πάνω να προέρχονται οι λύσεις. Όλες οι προτάσεις πάνε σε δημόσια διαβούλευση. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όλες τις ιδέες, να τις προωθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νάπολη. Αυτό για την Νάπολη είναι κάτι που μας ντροπιάζει όλους. Μας ντροπιάζει έτσι όπως τη διαχειριζόμαστε τόσα χρόνια. Δυστυχώς. Τα προβλήματα συσσωρεύονται και βρίσκαμε στη θέση πριν την οποία ακόμα και τις προτάσεις που λαμβάναμε κατέληγαν στο ότι ακόμα και τεφροτήρες θα πέραν 20 χρόνια για να κάνουν δουλειά. Άρα, να ασκηθεί πίεση να προχωρήσουμε καλύτερα. Όπω ξέρετε έχουμε και αυτό το... Τι αυτή επιστολή του 260, την επίσημη, το επίσημο διάβημα Προ τι ιστορικέ αρχέ, Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί συνέχεια η αυτήν, γιατί χρειαζόμαστε λύσεις. Ακόμα και αν λύσεις αυτές είναι πολύ πολύπλοκες. Ακόμα και όταν κάποιες λύσεις επιδέχονται βελτίωση, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γιατί κανείς δεν θα πρέπει να, την, να μην την ε, μετέλθει. Πολλές φορές είναι δύσκολο τα πράγματα, αλλά θα πρέπει κανείς από κάπου να ξεκινήσει και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ το στο εξής. Επομένως, μπορείτε να υπολογίζετε ότι εμείς αυτό θα κάνουμε. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να επιταχύνουμε την άνοιξη δράση Εμείς έχουμε τους τρόπους να το κάνουμε αυτό. Βέβαια έχουμε και τις εξαιρετικές περιστάσεις και με επιτυχία χρησιμοποίησαμε αυτή τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Δύο φορές το κάναμε αυτό με Ιταλία και Μάλτα για, ε, με την Πολωνία για, για τους Βέβαια αυτό μπορεί να γίνει με κάθε αναφορά. πολλές φορές, έχουμε κάποιες καταγγελίες. Πολλές φορές ήδη έχει γίνει ζημιά. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό και στις προτάσεις, στις συζητήσεις, όπως σας είπα σε μεκτήρες δηλώσεις μου, σας είπα τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Έτσι θα προχωρήσουμε. Να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε την οργάνωσή μας. Έτσι επομένω, θα δούμε πώς θα βελτιώσουμε το αυτό που ξέρουμε και όλοι να είμαστε καλύτεροι, καλύτεροι όσον αφορά όλες τις καταστάσεις από τις να τις αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Τώρα, αυτό η παρακολούθηση και τι γίνεται με τις κίτρινες αναφορέ. Ε, αναφορές. Βεβαίως και είναι σημαντική η παρακολούθηση. Καλά τα είπατε. Δεν, δεν, δεν έχω πρόβλημα. Κυρία Άκεν, σύμβαση του Άρχους. Το 2003, τότε που είχαμε αυτόν τον πυλώνα προς συζήτηση, ίσιαν άλλα από ό,τι σήμερα. Στο μεταξύ. Πέρασε συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε το χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων, είναι όλα ξεκάθαρα. Έχουμε ξεκάθαρη απόφαση του δικαστηρίου. Λένε ότι δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμη η σύμβαση του άρχους, άρα χρειάζεται εφαρμοστική νομοθεσία και γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε βάσιμους λόγους να αναθεωρήσουμε και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που είναι συγγενές με όσα ίσχυαν το 2003. διαφάνεια τώρα. Βεβαίως και είμαι υπέρ της διαφάνειας. Ξέρω όμως ότι αυτό είναι παλαιό αίτημα του Κοινοβουλίου. Και οι διατάξεις σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραβάσεις θα πρέπει να είναι ακριβώς όπως γίνεται και με όλους τους τομείς της πολιτικής. Οπότε, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Και έτσι θα βρούμε κάποιους, ε, κάποιες λύσεις. Προσπαθούμε κάποια θέματα να αντιμετωπίσουμε οριζόντια, εγκάρσια, αλλά δεν είναι πάντοτε αυτό εύκολο. Πάντω νομίζω ότι το... ο χρόνο είναι με το μέρο. Και έτσι ελπίζω ότι ισχύει. Τώρα για του αποτεφρωτήρε. Είναι σωστό αυτό που υπόθηκε. Και η κυρία Μάρκες ασχολείται με αυτό. Για, σχετικά με τα απόβλητα. Α, ξέχασα χθε να σας πω κάτι. Στο έγγραφό μας για τη σωστή χρήση των πόρων έχουμε σαν σκοπό να εγκαταλείψουμε τις χωματερές μέχρι το 2020. Προς τα εκεί κινούμαστε. Πρέπει να προσέξουμε όμως να μην πιέσουμε πολύ για την καύση. δεν ξέρω αν είναι εξίσου κακή η λύση οι καύσεις όπως ε, και οι χωματερέ, αλλά θα πρέπει να έχουμε σωστή ιεράρχηση. Λιγότερα απόβλητα θέλουμε, ανακύκλωση, επαναχρή, εκ νέου χρήση των αποβλήτων, ε, τελευταία η Είναι πρόσφατη προσέγγιση. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να μας ε, πούν πώς τα έχουν λάβει αυτά υπόψη. Πρέπει η ανακύκλωση να προωθηθεί, η εκ νέου χρήση κάποιων αποβλήτων. Η αποτέφρωση είναι καλή σε κάποιες ε, περιπτώσεις, αλλά δεν θα επικρατεί, δεν πρέπει να επικρατεί όσον αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων. Ε, Natura 2000 και η χρηματοδότηση αυτής. Νομίζω ότι στην αρχή εξήγησα το όλο θέμα. Η υποχρέωση να παρουσιαστούν εναλλακτικά προγράμματα. Ναι, αποτελεί ένα τμήμα της νομοθεσίας που Προσπαθούμε πάντα να εφαρμόζουμε και πάντα το ζητούμε. Όταν εξετάζουμε την ατούρα, αυτή είναι μία από τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Τώρα αν ικανοποιούμεθα με την απάντηση που δίδουν τα κράτη-μέλη είναι διαφορετικό θέμα. Πάντα επιμένουμε να εφαρμόζεται αυτή η αυστηρή λογική. Δηλαδή, οικονομικά συμφέροντα, κοινωνικά συμφέροντα πρώτα. Δεύτερον, να αποδειχθεί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Τρίτον, μέτρα αποζημίωσης, τα οποία αξιολογούμε από κοινού. Και αυτά τα μέτρα θα πρέπει, η αποζημίωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την απώλεια. Αυτό είναι και το νόημα της αποζημίωσης. Κλίμα, βιοπικιλότητα, συμφωνώ. Χρειάζεται προσέγγιση που λαμβάνει τα πάντα υπόψη. Συστηματική προσέγγιση. και το βασικό στοιχείο είναι η μακροχρόνια βιωσιμότητα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λύση άσπρο ή μαύρο. Πάντα στο τέλος πρέπει να κρίνει κανείς αν κάτι είναι ωφελές ή όχι. Ας πούμε το, τα ύδατα, ενέργεια από το νερό κλπ. Η χρήση της πράσινης ενέργειας κλπ. Όλα τα στοιχεία επαναλαμβάνονται υπόψη. Χρειάζεται σοβαρή ανάλυση επίσης. Τέλος. Regions of regions should yeah I I think that the voice of the voice from bottom up should absolutely be πρέπει να ακούγεται η επιτόπια φωνή, η προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, οι εταιρικές συμφωνίες σημαντικές για την υποστήριξη των περιφερειών και της βιωσιμότητας, σωστή προσέγγιση και για μας και για, τις, για την τοπική αυτοδίκηση. Εμείς και οι υπηρεσίες μας είμαστε συνεχή επαφή με τους αρμοδίους όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτή είναι η αιρεσιμότητα λοιπόν και είναι η συνήθις διαδικασία. Απαγόρευση των χωματερών. Εδώ κλείνω. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Ευχαριστώ Επίτροπε Ποτόρσνικ. Νομίζω ότι ήταν μια μέρα καρποφόρα για όλους μας. Μεταξύ άλλων μια συζήτηση που μας οδηγεί σε περαιτέρω δεσμεύσεις. Επιστρέφω στο βασικό θέμα. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα και ένα αίτημα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πείτε μου πώς να βελτιώσουμε τη συνεργασία. Αυτό είπε. Πρέπει να φανταστούμε σαφή συγκεκριμένη πρόταση να διατυπώσουμε προ τον Επίτροπο για να βελτιωθεί η συνεργασία μα. Λοιπόν, ευχαριστώ πραγματικά για τη συμμετοχή σα, για τη συνεισφορά σα που ήταν σημαντική. Sì, aspetta un attimo. Please, co colleagues, can you please take place? Ε, καθίστε, συνάδελφοι. So we can restart, okay? Allora, andiamo. Λοιπόν, εντάχει, πάμε στα επόμενα σημεία της ημερήσιας ε, διάταξης. Έχουμε την αφορά 551 Μίχα Ρεγκακάρ του Μίγκα Μίχα Ρεγκαχάρ, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτή την αναφορά δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Θα δώσω το λόγο στον Βίλιαμ Φλόιτ. λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πρόσφατη αυτή η αναφορά που προσθέθηκε εδώ στην Ινδοσία Διάταξη. Είναι σλοβενική ε, αναφορά και πήραν μια γραπτή ανακοίνωση από εμάς. Θα σας πω δύο λόγια για το, τι έχουμε να πούμε για αυτή την αναφορά, αν θέλετε. Αφορά δύο σημαντικά θέματα της, των οργανώσεων αυτών στη Το ένα είναι γνωστό, είναι το θέμα πλουσίων ε, αλλοδαπών που έρχονται στην αγορά ακινήτων σε μια χώρα που δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την εισβολή και το δεύτερο αφορά την προστασία μνημείων παγκοσμίου κληρονομιάς. Για το πρώτο σημείο, παρόλο ότι η σύσταση να αγνοηθεί αυτό το σημείο, είναι αρκετά σημαντικό. Το ξέρετε από παλιότερε ε, αναφορέ. Τα νέα κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν να οριστούν περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων μετά την ένταξή τους να περιοριστεί η είσοδος ε, αλλοδαπού κεφαλαίου στην αγορά κινήτων. Θυμόσαστε ίσως ε, την περίπτωση ενός Γερμανού αναφέροντος που ήθελε να αγοράσει στην Ουγγαρία ε, ένα αγρόκτημα και δεν μπορούσε γιατί η Ουγγαρία είχε ζητήσει παράταση αυτού του περιορισμού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον η Σλοβανία είχε ζητήσει μια τέτοια παρέκκληση ή όχι, αλλά μπορούμε να το λέξουμε και να το πούμε. Παρ' όλα αυτά θυμόσαστε στους κάποιες Ιλλανδικές ε, αναφορές, γιατί και στην Ολλανδία είχαν ένα πρόβλημα ε, έκρηξης της ε, αγοράς ακινητών, ξεδίες οποίες δεν μπορούσαν να, αγοράσουν οι ντόπιοι πια σπίτια και αναγκαστήκαμε να τους μιλήσουμε γιατί εν μέρη εξ αυτού είχαν αρχίσει να περιορίζουν ε, την ελευθερία εγκατάστασης. Αυτά μπορούν να γίνουν εφόσον είναι νόμιμος ο στόχος ε, των προσπαθειών. Το δεύτερο Ε, τμήμα ε, είναι κάπως αφήσει η αναφορά. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ε, λεπτομέρειες του αναφέροντος, το τι θέλει ακριβώς. Είναι αληθές ότι στην Σλοβονία το θέμα στραφοδότησης με είδωρ είμαστε πολύ καλά, 89% αλλά όσον αφορά την επεξεργασία των λιμάτων δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε καλό επίπεδο. Και υπάρχουν ορισμένε περιφέρειες όπου είναι πολύ ε, λεπτή η κατάσταση. Από το Ταμείο Συνοχής ε, ε, δαπανούνται κάπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την επεξεργασία των λιμάτων και μπορούμε να σας ενημερώσουμε τι γίνεται ακριβώς. Αλλά αυτά θα υποβληθούν αργότερα και θα ήθελα να σας ενθαρρύνουμε να έχουμε τον συγκεκριμένες λεπτομέρειες από τους αναφέροντες για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Ο συνάδελφος Γιάρ. Da stimmt dem zu. Ich würde nur noch die Anregung geben wollen. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ήθελα να πω το εξή. Για το πρώτο θέμα, το θέμα του αλλοδαπού κεφαλαίου στην ε, τόπια αγορά κινητών. Από ό,τι κατάλαβα αυτή η απόφαση, κατά πόσον ε, θα δοθούν ξαιρέσει ή όχι, είναι μια απόφαση του κράτους μέλους. Δεν αποφασίζεται εδώ δηλαδή. Θα πρέπει να το πούμε λοιπόν στον αναφερόμενο ότι το κράτος μέλος θα αποφασίσει αν κατάλαβα καλά, αν θέλει κάτι τέτοιο ή όχι. Εάν εμεί ω Επιτροπή Αναφορά θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι καλό και το πιστεύει και η Κομισιόν, θα πρέπει εκεί πέρα να περάσει στα χέρια του κράτου μέλου. Θα πρέπει να το πούμε αυτό στον αναφέροντα. Να στραφεί παραδείγματο χάρη στην Εθνική του Επιτροπή Αναφορά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη τη Σλοβενική κυβέρνηση. Αν δεν θέλει να παρατείνει την εξαίρεση αυτή, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αν κατάλαβα καλά. Non ci sono altri interventi? Δεν ζητάει άλλο το λόγο. Sicuramente c'è eh, Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες, αυτό είναι σίγουρο και για ευάθυνση. Το τόνισε αυτό και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως οι αναφέροντες μπορούν να δώσουν συμπληρωματικά στοιχεία. Καλό θα ήταν να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η αναφορά, να ζητήσουμε και άλλες πληροφορίες, να προβούμε σε μια επαφή, να έχουμε επαφή με την Επιτροπή για περισσότερες πληροφορίες και να πάρουμε μια απάντηση που θα είναι χρήσιμη για την υπόθεση που εξετάζει η Επιτροπή μας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, κλείνουμε αυτό το σημείο με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την αναφορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσει. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η αναφορά στο σημείο 18. Αντών Εντώνη και Ματία Ντοναντέλ, υπαριθμόν 804, δεν είναι παρόντε οι αναφέροντε. Θα δώσω αμέσω το λόγο λοιπόν στον υπεύθυνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Τζόναθαν Πάρκερ, δυνατό λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η περιφέρεια γύρω από την ε, Μέστρε είχε συμφόρηση κυκλοφορική και γι' αυτό άνοιξε ένας περιφερειακός ε, ε, το, η αναφορά θύχει τέσσερα συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν ότι το, θέμα, το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε και με διόδια που δεν προβλέπονται στο αρχικό ε, προσχέδιο. Δεύτερον, ότι δεν συμφωνώ με το Veneto City και το Ρωμαίο Κομερσιάλε. Τρίτον, ότι η συμφωνία για το ταπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τύχη σεβασμού και ε, κατά πόσον υπήρχε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πρώτο σημείο, η Κομισιόν δεν βρήκε να υπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το, το διαμόρφωση του οποίου δεν είναι νομοθεσία της, ενώ δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Κατά δεύτερα τα άλλα θέματα ζήτησε η Κομισιόν πληροφορίες από τις Ιταλικές Αρχές και πήρε αναλυτικές πληροφορίες που ήταν ικανοποιητικέ για την Κομισιόν και που υπευλήθη στην απάντησή μας Μαΐου 2011 προς την Επιτροπή Αναφορών. Δεν θα επαναλάβω όλα αυτά αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή για την ΜΕΣΤΡΕ προετοίμασε ένα καινούριο προκαταρτικό σχέδιο για δύο από τους σταθμούς διοδίων. Όπως ξέρουμε αυτή η διαδικασία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τις δύο εμπορικές ε, το ΜΕΑ Κομισάλε είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου ε, σχεδίου αυτοκινητοδρόμων Κατά το Veneto City είναι ένα πρόγραμμα, συμφωνία, ένα κόρτο του προγράμμα στην Ιταλία. Η πραγματική σημασία υποβρέθηκε σε διαδικασία ελέγχου βάση οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Και αυτό εγκατακλείδη. Πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία ελέγχου της περιβαλλοντικής εκτίμησης Δεύτερον, δύο παρόμοιες ε, διαδικασίες προχωρούν και μία προγραμματική έχει ήδη λάβει χώρα. Δεν βλέπω λοιπόν καταπάτηση της κοινοτική νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ζητεί κάποιο συνάδελφο το λόγο. Όσον αφορά λοιπόν το σημείο λαμβάνοντα υπόψη την απάντηση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να αποφασίσουμε να κλείσει η συγκεκριμένη αναφορά διότι ήταν εξαντλητική αυτή η ανακοίνωση. Ίσως μπορούν οι αναφέροντες να επαληθεύσουν τι γίνεται το νέο πρόγραμμα και τι βήματα θα ακολουθήσουν. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την αναφορά και πάμε στο επόμενο σημείο. Ε, είναι οι αναφορές που είναι στο σημείο 19 που υπευλήθησαν από τον κύριο Ρομπέρτο Τζουραστάντε αφορούν το ίδιο θέμα και σε αυτή την περίπτωση. Α, τρεις είναι οι αναφορές ζητού, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, που συζητούνται από κοινού, διότι αφορούν το ίδιο θέμα. Και εδώ δεν έχουμε τους αναφέροντες, τον αναφέροντα, τους αναφέροντες μάλλον παρόντες. Δίνουμε το λόγο στην υπεύθυνο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στην κυρία Μπελίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εξολόγηση αυτών των ε, αναφορών οδήγησε σε πολλές γραπτές ε, ανακοινώσεις. Και ο Επίτροπος Ποτόσνικ έκανε κάποιες ε, παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Όσον αφορά το σχέδιο αυτό για την Τριέστη, για την επανειλοποίηση, δεν έχει δοθεί ακόμα η σχετική άδεια βάσει των πληροφοριών που ε, λήφθησαν από τις Ιταλικές αρχές και που υποβλήθηκαν από τους αναφέροντες, η Κομισιόν δεν βρήκε να υπάρχει καταπάτηση της κοινωτικής νομοθεσίας όσον αφορά αυτέ τι μονάδε επανειριοποίηση κοντά στον κόλπο τη Επίση, η αναφορά αυτή αφορά την εφαρμογή του άρθρου 131 τη οδηγία Σεβέζο στην Τεριέστη. Η Κομισιόν ε, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των απαντήσεων που εδόθησαν από την Ιταλική κυβέρνηση για το θέμα και αποφάσισε να εκτώσει προειδοποιητική επιστολή κατά της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 2010. Οι Ιταλικές αρχές τώρα ε, θέλουν να συμμορφωθούν με τι διατάξει τη Συμφωνίας του Εβέζο όσον αφορά την ε, συμπεριφορά σε περίπτωση του Συγκεκριμένα, για το άρθρο 13.1 οι αρμοδιότητες είναι στη Σάββατη Βαρδαβάνα, Βούτα και Τριέστε. Οι Ιταλικέ αρχέ ενημέρωσαν την Κομισιόν για μια σειρά πρωτοβουλειών που υιοθέτησαν για να εξασφαλίσουν την ενημέρωση του πληθυσμού που αφοράται ίσω σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματο από την εγκατάσταση αυτή. Αυτέ οι πρωτοβουλίε σημαίνει ότι διατίθεται η πληροφορία αυτή μέσω διαδικτύου. Ε, Πληροφορίε που θα πρέπει να έχουν δοθεί εκ των προτέρων όσον αφορά την συμπεριφορά σε περίπτωση ε, δυστυχήματο, βάσει δηλαδή της οδηγίας ΕΒΕΖΟ και επίσης η ενημέρωση των λογομονάδων σε περίπτωση δυστυχήματο. Και στείλαμε τι σχετικέ πληροφορίε στον αναφέροντα για να τον ενημερώσουμε για το περιεχόμενο της απάντηση Ιταλία και για το γεγονό ότι οι υπηρεσίε Κομισιόν θεωρούν θετικά αυτές τις απαντήσει Η Κομισιόν θα κρατήσει ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για οποιοδήποτε θα εξελίξει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σύντομο σχόλιο έχω όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιλώ Ιταλικά αυτή τη φορά διότι είχα την ευκαιρία επανειλημμένα να συναντηθώ με τους εκπροσώπους της οργανώσεως ε, των, πολιτών στο, στην Τεργέστη και θαύμασα πώς αυτές οι οργανώσεις μπορούν να μιλούν για πραγματικά προβλήματα και πώς είναι σε θέση να συνεννοούνται και να καταλήγουν κάπου σε κάποια λύση όσον αφορά το πρόβλημα που συζητούν. Αυτές οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το είπα και παρουσία του Επιτρόπου Ποτότσνικ αυτό. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τη λογική του θεματοφύλακα των συνθήκων. Όμως ένας παθητικός θεματοφύλαξ. Είναι σαν να μη συνέβη τίποτα, είναι επικίνδυνο όμως το παιχνίδι, ίσως κάτι να συμβεί, έτσι ακούγονται με αυτά που λένε. Όμως για την ώρα είμαστε σε ασφαλές έδαφος. Χρειάζεται, πιστεύω, λίγο πιο συγκεκριμένη η γλώσσα. Πρέπει να ακούσετε τα επιχειρήματα των περιβαλλοντικών οργανώσεων παρά την απουσία τους. Δεν είναι παρόντες γιατί είναι δύσκολο να έρθουν. Ενώ για τις επιχειρήσεις είναι πιο εύκολο γιατί έχουν χρήματα αισθάνομαι καθήκον μου να εκπροσωπήσω τη φωνή τους και περιμένω σαφέστερη τοποθέτηση, πιο αποφασιστική στάση, πιο ανοιχτή από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μιλάμε για αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Μπεγιέρ. Je vais aller dans le sens euh, de ce qu'a énoncé mon collègue. Parce... που είπε ο συνάδελφος. Δεν είναι πολύ σαφής η κατάσταση σε αυτή την εξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει κάποιες σκιές. Τι λέει η Ιταλία, τι εγγύες υπάρχουν. Υπάρχει έγκριση για αυτά τα έργα, προγράμματα. Τι γίνεται με την ομοθεσία για αυτά τα επικίνδυνα έργα. Θα πρέπει να μην υπάρχει και αμφιβολίες για τέτοια θέματα. Άρα, εγώ προτείνω να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά, ούτως ώστε να συνεχιστεί ο διάλογο. Και να συνεχίσουμε να ασκούμε την αποδοτική πίεση. Πέτερλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω μετάφραση προς τα σλοβενικά και θα μιλήσω στα αγγλικά. Έλαβα μια σειρά επιστολών σε σχέση με αυτή την ε, αναφορά για το θέμα αυτό. Έχω σχοληθεί με το περιβάλλον από υπεύθυνες θέσει στη χώρα μου και ξέρω πόσο λεπτό ευαίσθητο θέμα είναι το περιβάλλον. Και επίσης συμμερίζομαι τον προβληματισμό του κόσμου και των διαφορών φορέων όσον αφορά το μέλλον. Έκο, Γιατί εδώ υπάρχουν συγκεκριμένε ε, απειλέ που αναδύονται γι' αυτό και είναι σημαντικό ο κόσμο να ξέρει ότι υπάρχουν κανόνες και ότι εφαρμόζονται. Και συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος Βάγκελ. Ότι δηλαδή είναι σημαντικό ο κόσμος να διαπιστώνει το ότι ενδιαφέρεται η Κομισιόν στρατεύεται, ας το πούμε. Να υπολογίζουν στο ότι η Κομισιόν ή η ΟΚ θα προσέξει το θέμα. Επίση προβληματίζομαι Λέω ο ότι δεν είναι βέβαιος ότι υπάρχει ενημέρωση για τις επιπτώσεις εκεί, σε, αυτό το, σε αυτή την περιοχή τη Ευρώπης. επομένω, ήδη το ότι γίνονται όσα γίνονται είναι πάρα πολύ θετικό. Ελπίζω δεν έχουμε εδώ να κάνουμε εκτελεσμένα και όσον αφορά τη συνέχεια της διαδρομής είναι σημαντικό ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχει επαρκής ενημέρωση. και εγώ ότι υπάρχει τήρηση της νομοθεσίας. Επομένως, προς τα εκεί ελπίζω ότι θα πάνε τα πράγματα. Επίσης, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν έχουμε εδώ το κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες για τέτοιου είδου ε, επενδύσεις. Ε, πρόκειται εδώ πέρα για τρεις διαφορετικές χώρες. Ευχαριστώ. Γεια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, γιατί και η ίδια Κομισιόν ε, λέει στο κείμενο ανοιχτά ότι οι Ιταλικές Αρχές θα έχουν δώσει λεπτομερείς ε, πληροφορίες για κάποιες εγκαταστάσεις στην εταιρεία και οι πληροφορίες αυτές ε, επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες της Κομισιόν. Θα πρέπει να γίνει εις βάθος και γλίγορη εξέταση, ούτως ώστε να μπορούσαμε εμείς στην Επιτροπή Αναφορά του Λιγοράτου Δυνατών να ξαναεξτάσουμε αυτήν την αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Η αναφορά παραμένει λοιπόν ανοιχτή και θα τη συζητήσουμε ακολούθως αργότερα όταν θα έχουμε και άλλες πληροφορίες για να καθορίσουμε θέση μας. Ευχαριστώ. Περνώ στην αναφορά του σημείου 20. Είναι εδώ παρόντες οι αναφέροντες. Ο κύριος Ζαν Φιλίπ Γκαλόν εκπροσωπεί την Ένωση και του δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Madame la Présidente, euh, Mesdames, Messieurs les Parlementaires, nous Λοιπόν, κύριοι, κυρίες βουλευτές, ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε ξανά τη βοήθειά σας. Εδώ και μερικούς μήνες δύο συνάδελφοι σας μίλησαν για το σχέδιο κενήτων που είναι κοντά στην παράκτια περιοχή σε παλιές ε, λόγες λασπόδης περιοχές. εγκαταλήφθηκε το σχέδιο έκτοτε και σήμερα θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θερμά γι' αυτό. Ε, μαζί μας φέραμε ένα, κάποιες διαφάνειες. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εκεί μεταξύ Γκεράν και Μπάσιρ Μέρ Έχουμε 1.800 εκτάρια θαλασσινού νερού και είναι από τα θαύματα αλμυρού νερού και είναι θαύματα της Βρετάνης και της Δυτικής Ευρώπης, θα έλεγα, είναι ένα θαύμα. Λοιπόν, βλέπετε ότι βγαίνει στη θάλασσα το έδαφος και έχουμε εκεί πέρα τους κατοίκους που καλλιεργούν, αν θέλετε, τις περιοχές αυτές κοντά στον ε, Ατλαντικό και ε, καλλιεργούν τα χωράφια τους με γεωμετρικό τρόπο και βλέπετε είναι ένα μοναδικό τοπίο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Λοιπόν, είναι παράξενο το εδαφός χωρίς δέντρα, ε, περπατάει κανείς ε, σαν τους Ασιάτες ε, που περπατάνε στους οριζόνες, αυτό θυμίζει. Λοιπόν, δεν βάζουν λιπάσματα, δεν βάζουν παρασιτοκτόνα, δεν βάζουν γεωργικούς ελκυστήρες εκεί. Λοιπόν, οι καλλιεργητές εκεί χρησιμοποιούν τεχνολογία την πιο ήπια που υπάρχει, κόβοντας με το χέρι, μαζεύοντας με το χέρι το αλάτι και τον καρπό του αλατιού. Ε, τα σχήματα που χρησιμοποιούνται είναι ενέργεια που συλλέγεται από τον άνεμο, τον ήλιο και τη θάλασσα και από το θαλασσινό νερό. Λοιπόν, αυτά τα υφάλμυρα νερά είναι οικολογικός ε, πλούτος. Ε, και ε, εδώ και αιώνες οι καλλιεργητές εκεί διασφαλίζουν τη διόνυσή τους. Ε, Υπάρχουν πάρα πολλά ζώα και φυτά εκεί πέρα, μεγάλη βιοπικιλότητα, την εγκαταλεύονται διάφορα είδη των θαλασσίων ειδών και των πτηνών ε, που μένουν εκεί, είτε είναι μετανασταυτικά τα ζώα και τα πουλιά, είτε μένουν εκεί. 180 είδη πτηνών έχουν καταγραφεί, 159 είναι μόνιμα είδη που μένουν εκεί 72 εκεί έχουν τις φωλιές τους ε, είναι, πολλά, είναι 7 πολύ σπάνια είδη και 8 πάρα πολύ σπάνια και στη Γαλλία και στην Ευρώπη από όλα αυτά τα πουλιά 12 από αυτά τα φυτά, α, ε, συγγνώμη, τα ζώα αυτά αναφέρονται στα διεθνή ε, κείμενα που αφορούν την προστασία των περιοχών στα οποία ζουν αυτά τα ζώα. Λοιπόν, εδώ, σε αυτή τη χερσόνησο μεταξύ ωκεανού και υφάλμηρου ύδατος, στο Πουλγκό, στην περιοχή του Πουλγκό, σε περιοχή Natura 2000, σε ταξινομημένη περιοχή. Ε, λοιπόν, εκεί, ε, εδώ και πολλά χρόνια ε, υπάρχουν διάφοροι ε, κάτοικοι. Υπάρχουν ζώνες όπου τρέφονται τα ζώα, εκεί πέρα. υπάρχουν ύβιδες, υπάρχουν, υπάρχει ύβης, υπάρχουν διάφορα ζώα και είναι αξιοσημείωτα θέαμα και είναι θέαμα, θεαματικό το θέαμα των ζώων που μαζεύονται εκεί. Όπως βλέπετε. Να και μια είδηση. Λοιπόν, κλασική εξέλιξη αυτή για αυτά τα πουλιά. 20 φόλιε ε, απαριθμήθηκαν από την άνοιξη του 2010 και οι ντόπιοι ορθινηθολόγοι το επιβεβαιώνουν και φέτος. Σήμερα αυτά τα ίδια απειλούνται όμως. τον Ιούνιο του 2010 μη αδειοδοτημένες εργασίες κατέστρεψαν αυτό το τοπίο. Αυτό το κόκκινο κομμάτι είναι κοντά στο δάσος που επιτρέπει το να ε, πηγαίνουν τα πτηνά και έχουν χαθεί πρόκειται για σκόπιμης ε, προσπάθειας που έγινε εκεί πέρα Ορίστε οι εργασίες που έγιναν που επηρέασαν, έπληξαν τις φωλιές των πουλιών. Μια επιχείρηση το έκανε αυτό. Ε, διευθυντής είναι και ερετός, πρώην δήμαρχος που συμμετείχε στην, ε, στον καθορισμό της περιοχής Ανατούρα 2000 αλλά είναι σκόπιμη αυτή η προσέγγιση χωρίς κινδύνους, ατιμωρητή Κανείς δεν ζήτησε την επιβολή υποδειγματικών ποινών ούτως ώστε ε, όταν καθορίζεται με περιοχή ε, Natura 2000 να το σκέφτονται δύο φορές όσοι θέλουν να προσβάλλουν τις συγκεκριμένες περιοχές. Και σας λέμε σήμερα, είμαστε μπροστά σας και σας λέμε πρέπει να μας βοηθήσετε, συνέβησαν αυτά τα πράγματα, να τι συμβαίνει, να τι θα συμβεί. Πάντα υπήρχαν αυτά τα ζώα εκεί πέρα. Εδώ είναι η τοποθεσία όταν αποκαταστάθηκε, αλλά δεν θέλαμε αυτό το αποτέλεσμα την αποκατάσταση. Γιατί. Βλέπουμε τη περιοχή Natura 2000 στα γαλάζια, κόκκινο, βλέπουμε το έργο που είναι προσιλοποίηση. Κινούνται γρήγορα, δεν τους νοιάζει τι καταστρέφουν. Θέλουν να μειώσουν και την περιοχή και τη ζώνη Natura 2000 Αυτό είναι το σχέδιο αυτό το στοιχό που εφαρμόζεται. Βλέπετε το, το κομμάτι με τα προστατευμένα ήδη εκεί στο τέλος του βέλους. Έπρεπε να απέχουν τουλάχιστον από, τα, από την πανίδα ε, τουλάχιστον 30 μέτρα. Υπάρχει και δρόμος κατασκευή επίσης. Αυτά. Είναι τετελεσμένο γεγονός αυτά τα οικοδομήματα παράνομη κατασκευή σε Natura 2000. Και η χώρα, το κράτος δεν τιμωρεί αυτούς παραβίασαν. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εφαρμογή υποδειγματικών κυρώσεων για να είναι αποτρεπτικά τα μέτρα στο μέλλον. Διαφορετικά θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Si Να προσθέσω κάτι. Ότι έχουμε, κάνει, έχουμε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα τον εισαγγελέα. Και απορρίφθη το αίτημά μας. Ε, αυτός που διαπράττει την παρανομία είναι πρώην δήμαρχος και ίσως δεν ξέρω, δεν είναι κάποιος ξένος. Ευχαριστώ. Στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιστροπής, Ζόζεφ Βάντερ Στίγκεν, δίνω το λόγο. Oui, Madame la Présidente. Merci. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να συνοψίσουμε το τι έγινε όπως έκανε ο προλαλής σας. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές ε, αλλαγές όσον αφορά αυτό το εδάφιο για αυτή την ειδική προστατευμένη περιοχή σε αυτό τον ε, βαλτότοπο. Έγιναν επομένως κάποιες παρεμβάσεις και έχουμε τώρα δύο καταγγελίες. Πρώτα-πρώτα λέω αναφερομένως ότι εδώ υπήρξε αλλίωση του περιβάλλοντος και ότι σταμάτησε να προστατεύονται τα πουλιά. Και άρα υπάρχει παραβίαση της οδηγίας του περιβάλλον. Επίσης εδώ καταγγέλλεται η χωροταξία γιατί εκεί πέρα υπάρχουν παραδοσιακές δραστηριότητε και, και αυτό επίσης ε, λέει ότι δεν είναι σωστό όσον αφορά την, το, το περιβάλλον. Και τώρα πάμε στο άρθρο 6 παραγωγός 3 της σχετικής για το περιβάλλον ε, και οπότε ε, εδώ είναι δυνατόν να έχουμε μία αξιολόγηση που θα πρέπει να γίνει για το τι έγινε και για το πόσο υπάρχει προστασία αυτού του χώρου. Το Natura 2000 δεν αποκλείει οποιαδήποτε παρέμβαση για ανοικοδόμηση. Θα πρέπει όμως να τηρούνται οι διατάξεις της τρίτης και τέταρτης παραγράφου του άρθρου 6. Επομένως, εμείς πού καταλήγουμε όσον αφορά τις αλλοιώσεις για αυτή την, τον καθαρισμό. Οπότε θα πρέπει να επαναφέρουν τα πράγματα και όπως ήταν. Το δάσος είναι, το δάσος είναι ε, άθικτο και δεν θεωρούμε ότι έχουν παραβλαβεί τόσο πολύ τα πουλιά. Ευχαριστούμε για τις όσες πληροφορίες μας έδωσε ο αναφερόμενος και όσον αφορά την τροποποίηση του τοπικού σχεδίου χωροταξίας θεωρούμε ότι ούτε εδώ υπάρχει ασυμβατότης με το Natura 2000. Όμως θα πρέπει να γίνει προηγουμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων, να δούμε αν υπάρχει σημαντική επίπτωση. Και για το μέλλον επομένως το τι θα γίνει πλέον ταξικής θα εξαρτάται από αυτά που προείπαμε. Θα πρέπει να γίνει επομένως αξιολόγηση περιβαλλοντική επί τη βάση του τοπικού προγράμματος ανοικοδόμησης και χωροταξίας και θα πρέπει να δούμε αν έγινε αυτό και κατά πόσον θα υπάρχει τώρα σημαντική επίπτωση όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον και την τοπική πανίδα σε σχέση με το Natura 2000. Απευθυνθήκαμε στις γαλλικές αρχές και είπαμε ότι θέλουμε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με το πώς εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από την χωροταξία που σχεδίασαν. Υπήρξαν πληροφορίες, θέλουμε κι άλλες. Βεβαίως και πρόκειται να σας ενημερώσουμε για την συνέχεια. Ευχαριστώ. Μπελιέ, συνάδελφος Μπελιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Δεν θα έχουμε πολλέ συζητήσει νομίζω για το θέμα αυτό, γιατί η Κομισιόν ολοκλήρωσε την παρέμβασή τη λέγοντα ότι αναμένεται μία αίτηση για περαιτέρω μελέτη. Θα είναι λοιπόν δικαιολογημένο να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Παρ' αυτά θα ήθελα, το έκανα βέβαια αναφέροντα, θα ήθελα λίγο να υπενθυμίσω στου συναδέλφου και να αναρωτηθούν για το φάκελο αυτό που εξετάσαμε εδώ και δύο χρόνια. Υπήρχε ένα σχέδιο χωροταξία, ακυρώθηκε, τώρα έχουμε ένα άλλο σχέδιο διαφορετική ε, χωροταξία για τη ζώμη αυτή. Εσείς ε, μιλάτε για ζώνες ε, οι οποίες μπορούν εύκολα να, μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να κρίνουμε την συμβατότητα μεταξύ μιας ζώνης που είναι η Natura 2000 για την προστασία των ειδών και μια ζώνη για ε, μικρή τεχνική δραστηριότητα θα πρέπει να υπάρχει ναι. μία προστασία των ευαισθητών περιοχών της Natura 2000, αλλά δεν πρέπει να απορρίψουμε εκ των προτέρων ότι μπορεί να, δεχθούμε εκ παραλλήλου τη δυνατότητα της ανάπτυξης μικρών οικονομικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της ε, τοπικής χωροταξίας Μου φαίνεται δύσκολο να δεχθούμε σε τόσο ευαίσθητες ε, περιφέρειες όπως αυτή να δεχθούμε εκ των προτέρων την συμβατότητα μιας βιομηχανικής ε, ζώνης και μιας ε, ζώνης περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα ήταν καλό να έχουμε κάποιες ευκρινήσεις από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν αυτή τη στιγμή εναμονή όλων αυτών των ε, διευκρινήσεων μπορούσε νομίζω να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και εάν δεν γίνει αυτή τη στιγμή τίποτα, ε, θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη αναφορά. Νομίζω ότι η Γερόντ δεν αρκείται στην ποιότητα της φύσης που είναι αναγνωρισμένη τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα πολύ καλύτερα για το περιβάλλον εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ε, άλλες ε, παρεμβάσεις από πλευρά συνάδελφων. Συνάδελφος Μπολά. Πολύ σύντομα γιατί δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εδώ με τις ώρες. Το θέμα είναι αρκετά σαφές κατά τη γνώμη μου. Εκτός από ένα-δύο σημεία δεν κατάλαβα ποιο, ποιο ήταν η αιτιολόγηση της απόρριψης ε, της προσφυγής που υπέβαλε η, ε, η επιχείρησή σας. Επίσης, ποια ήταν η φύση των ε, αήλων βλαβών. Επίσης, κατά πόσον εδώ μπορούμε να έχουμε μια ζώνη δραστηριοτήτων που να είναι συμβατή με την ε, Natura 2000. Εγώ εκ των προτέρων δεν βλέπω κανένα μεγάλο πρόβλημα. Εσείς λέτε βέβαια ότι επειδή είναι ένας ερετός της τοπικής αυτοδίτησης εκείνος ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα με ναι, κρίνεται. Εγώ είμαι ερετός ε, στη τοπική μου περιφέρεια και δεν θεωρώ ότι είμαι υπεράνω των νόμων. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κανένας ε, σε επαγρύπνηση, αλλά δεν θα πρέπει να γυμνοποιούμε. Βέβαια, αυτές οι ζώνες πλήττονται με βιομηχανικές ε, ή χωροταξικές δραστηριότητες. Ή πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά, αναμένοντας όλες τις απαντήσεις και ιδίω την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης αξιολογικών ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Στην Αυτά γίνονται στη Γαλλία, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία απλή ερώτηση. Οι εργασίες του 2010 έγιναν χωρίς άδεια. Και στρέφουμε εδώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν αυτό είναι λεθές, είναι μια σαφής καταπάτηση της οδηγίας Natura 2000. Δεύτερον, Πού είναι οι εγγυήσει που αυτό το σχέδιο ε, για παραδοσιακές δραστηριότητες έχουν δοθεί. Πώς ξέρουμε ότι αυτό δεν θα μεταφερθεί, δεν θα μετατραπεί σε βιομηχανική δραστηριότητα. Αν δεν έχουμε εγγυήσει, γιατί να δεχθούμε αυτή την, αυτό το σκεπτικό του και σερά σερά ότι είναι να γίνει, θα γίνει δεν ξέρουμε στο μέλλον. Και επίσης η μελέτη της επίπτωσης παρέμβασης του ανθρώπου σε όλα τα ε, τμήματα της οδηγίας Natura 2000. Η οδηγία προβλέπει ότι αυτή η επίπτωση του ανθρώπου θα ελέγχεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για να αποφευχθούν οποιασδήποτε βλάβες. Έχουμε αυτές τις απαντήσεις σήμερα. Όχι, δεν τις έχουμε και γι' αυτό υποστηρίζω την ιδέα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και οι απαραίτητες εγγύησεις να προετοιμαστούν από τις γαλλικές αρχές. Και θέλω να πω και στο κύριο Βουλάρκ, τον Γάλλο φίλο μου, και σε άλλες χώρες που είναι επίσης μέση, μέλη της Ένωσης, επίσης δημοκρατικές χώρες, και υπό κράτος δικαίου αυτό λέγεται σύγκρουση συμφερόντων. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω δύο διευκρινήσεις, λέει κυρία Βουλή. Ιδίω έχω να ακούσει τον συνάδελφο Μπουλόμ. Ποια είναι η φύση των ε, απορριμμάτων αυτών που χρησιμοποιήθηκαν για τις προσχώσεις. Όποια και είναι αυτά, με σοκάρει ερώτηση, γιατί όποια και είναι αυτά, όσο επικίνδυνα ή μία επικίνδυνα είναι, είναι απαράδεκτο στην Ευρώπη να μπορέσει κανένας να επιτρέψει στον εαυτό του χωρίς άδεια, αφήνοντας καραμένος όλες τις ε, διαδικασίες που υπάρχουν για την αδειοδότηση, να ανοίξει μία τρύπα στον κήπο του και να βάλει μέσα ό,τι θέλει. Λοιπόν, για το θέμα αυτό, η φύση αυτών των ε, απορριμμάτων που χρησιμοποιήθηκε δεν παίζει κανένα ρόλο. Και θέλω να διευκρινίσω ότι στη Γαλλία όταν υπάρχει απλή προσφυγή, αν κατάλαβα καλά κάνατε μια τέτοια απλή προσφυγή, ο εισηγηλέας έχει την δυνατότητα να αποφασίσει αν θα δώσει συνεχή ή όχι. Αλλιώς ο δικαστής θα έπρεπε να δράσει και δεν θα είχε δυνατότητα επιλογής εάν η προσφυγή είχε υποβληθεί κάτω από διαφορετική, ε, διαφορετική μορφή. Αλλά όπως λέω αναφέρον, πραγματικά, στη Γαλλία όταν υποχρεούται η δικαιοσύνη να διώξει μια παράβαση κοστίζει σήμερα αυτό. Και ακόμα και στη ε, Γαλλία υπάρχουν άνθρωποι και ενώσεις που δεν έχουν τους πόρους για να μπορέσουν να προσφύγουν. Και αυτό μας κάνει να ε, επανέλθουμε στη σημασία του τρίτου, της τρίτης πτυχές ε, της σύμβασης, δηλαδή η δυνατότητα να έχουν οι πολίτες τα μέσα για να μπορούν να προσφύγουν για εργασίες τέτοιου τύπου στην ε, περιοχή τους. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Μπουλάν. Παρακαλώ, είστε σύντομοι. Διαφορετικά θα ολοκληρώσουμε. Θα είμαι πολύ σύντομο να πω σαν Τριμπελίξ. Αν αυτό το ερώτημα για το θέμα Natura 2000, είναι την προοπτική ενδεχομένη προσφυγή. Δεν κρίνω. Είναι εν ώψη προσφυγή όσον αφορά την φύση του, και τη ζημία που προκαλείται από αυτό για το περιβάλλον και την Natura 2000 γιατί βρίσκω λίγο υπερβολική την προσέγγιση παραγματική παράβαση συνέβη πρέπει να τιμωρηθεί είναι υπερβολικό όμως το ότι έγινε αυτή την προσφυγή δεν ποια ήταν η φύση της βλάβης. Μέσω μακροπρόθεσμα υπήρξαν βλάβες για το περιβάλλον ε, πέρα από το, αυτό που έγινε με τη μεταφορά των χωμάτων κλπ. Συνάδελφος Παλιαντέλη. Στην ε, Επιτροπή, ε, με αφορμή την τελευταία παράγραφο στο κείμενο που έχω στη διάθεσή μου, <clears throat> ότι η εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι η αποκατάσταση του τοπίου στη συγκεκριμένη περίπτωση έπειτα από την αφαίρεση του εδάφους εμπίπτει στην αρμοδιότητα των γαλλικών αρχών. Αναρωτιέμαι πού βρίσκεται η ευθύνη της, Ευ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την προστασία των ζωνών Natura 2000. Εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να υπερβούμε τα εθνικά όρια και να επιβάλλουμε πρόστιμα αφού παραβαίνονται όρια που έχουν ξεκαθαριστεί ότι είναι της Natura 2000. Πού βρίσκεται η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Μια απάντηση από την Επιτροπή. Η εφαρμογή της οδηγίας είναι για τους βιοτόπους και για τα πτήνα. Είναι ευθύνη της Γαλλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την εξουσία εκτός το να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αποδεδειγμένες υποθέσεις ε, αλλά είναι ευθύνη της χώρας. No, λίγα λεπτά να απαντήσει ε, αναφέρον. Ε, να απαντήσω συντομία στο ερώτημα που ετέθη από την κυρία Μπελιέ, τον κύριο Μπουλάν και άλλους. Ζητώ συγγνώμη τους άλλους τώρα αυτή η παραδοσιακή περιοχή δραστηριοτήτων, παραδοσιακών ε, δραστηριοτήτων, δεν βάλαμε διάφορες διαφάνειες πάνω σε αυτό, διότι μας ζητήθηκε να περιοριστούμε στο χρόνο που μας διατέθη. Θα μπορούσαμε να σας δείξουμε διάφορα εργαστήρια, τα οποία ήδη είχαν κατοικίες στον Άνω Όροφο, αρκετά σπίτια καινούρια, στριμωγμένα ανάμεσα σε δύο εμπορικά, εμπορικούς χώρους και στις φωτογραφίες είδατε ότι τεράστια αγορά είχε κατασταθεί στην ε, περίφημη αυτή περίπτωση. Τα εδάφια από τις προσχώσεις υπάρχουν διάφορα είδη, παλιά τούβλα υπήρχαν και, υπήρχαν και υπήρχε και αμύαντος ενδεχομένω. Τα άλλα ήταν ε, αδρανή απόβλητα, αλλά και κατάλοιπα ε, πίσας και λοιπά από πάρκιν, από κόρο πάρκιν. Για να απαντήσω τον κύριο Μπουλάνος, ο ερετός πρώην δήμαρχος και διευθυντής της επιχειρήσεως που είναι υπεύθυνη για τις εργασίες. Ε, έχει επαναλάβει το αδίκημα, ήδη το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν σε μια, στο ΣΕΜΟΛΦ, μια κοινότητα γειτονική, βάζοντας προσχώσεις αυτές σε ιδιωτικό κτήμα που δεν του ανήκε και χωρίς άδεια. Είχε, έγινε διαδήλωση των χωρικών και των τοπικών φορέων ε, και συνδικάτων. Γιατί ήρθαμε και γιατί μετακινηθήκαμε που κοστίζει χρήματα όπως έλεγε η κυρία Μπελίε για να σας ζητήσουμε αυτή η υπόθεση να τιμωρηθεί, να παραμείνει ανοιχτή και αν θέλετε είναι μια έκκληση για βοήθεια αυτή. Ο νομάρχης δήλωσε ότι είναι παράνομες αυτές οι εργασίες και γι' αυτό καταθέσαμε περιοριστική αυτή ε, καταγγελία. Τελικά δεν δόθηκε συνέχεια αυτού του είδους οι εργασίες δεν τιμωρούνται, δεν κυρώνονται σύμφωνα με το κείμενο Natura 2000 κλπ. Μας το είπε ο εισαγγελέα στο, στην αλληλογραφία του. Αλλά ο νομάρχης, τον οποίον ειδοποίησαμε από την αρχή των εργασιών, δήλωσε ότι αυτές οι εργασίες είναι παράνομες και γίνονται χωρίς άδεια σε τοποθεσία Natura 2000. Συμπέρασμα από εμά εξαρτιόταν από τις ορνηθολόγους της Ενώσης και λοιπά να κάνουμε τα διαβήματα και όπως έλεγε η κυρία Μπελιέ προβλέψαμε να προσφύγουμε στα αστικά δικαστήρια, αλλά πρέπει να πληρώσουμε τις δαπάνες και είναι σαφές ότι αν χάνουμε, όχι μόνο χα... χάνουμε την υπόθεση, αλλά πρέπει να πληρώσουμε ζημίες και, και τόκους. Μια άλλη οργάνωση ε, που έκανε το επέπαθε κάτι, έχασε την υπόθεση, είναι στα πρόθυρα της χειροκοπίας και δεν μπορεί να συνεχίσει την εργασία για προστασία της φύσης είναι μια οργάνωση για την προστασία των παρακτήων περιοχών. Ευχαριστώ, είναι μια έκκληση για βοήθεια. Αυτά ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, παραμένει ανοιχτή η αναφορά και μπορούμε να προσθέσουμε ότι περιμένουμε ήδη ε, κάποια άλλη ζητούμε από την τοπική, τοπικές αρχές ε, επιτάχυνση των ε, διαδικασιών να μας ταλούν τα έγγραφα ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε και να προχωρήσουν οι συζητήσεις ανάλογα με τις απαντήσεις που μας δοθούν. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που μας πρότειναν από το θέμα. Πάμε στην επόμενη αναφορά που είναι η 755 του 2010 του Τόνι Λόους. Είναι παρόν ο αναφέρον και στον οποίο δίνω το λόγο. Eh, eh, Σε δίνω κάποιο χρόνο έτσι για να τακτοποιηθείτε. Να ασχοληθούμε με την άλλη αναφορά το μεταξύ που δεν υπάρχει εδώ αναφέρον. Να κάνουμε παρουσίαση της επόμενης αναφοράς. Ενώ εσεί οργανώνόσαστε. Ωραία. Ah, no, it is... It's the final one. The... Subsequent Επόμενο θέμα είναι έκθεση της κυρίας Βάλεαν. No. Okay. You are... you ready? Okay. It's the same. Thank you, Chair, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη σημερινή μας αναφορά. Άντριο ονομάζομαι και προέρχομαι από τον ε, φορέα φίλη του περιβάλλοντος Ιρλανδίας και σχετικά με την εξόρυξη της τύρφης στην Ιρλανδία. Ε, έχουμε τρία σημεία να σας τονίσουμε. Το πρώτο είναι η σχέση μας με την τύρφη. Εκμετάλλευση γίνεται. Καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν έχω καταφέρει να εφαρμόσω την αυτοκινητικό μου. Ούτε στις προσταθόμενες ούτε στις άλλες περιοχές. Τίποτα δεν γίνεται με το κεκτημένο. Και ο λόγος που ήρθαμε σήμερα εδώ είναι να σας δείξουμε τι ισχύει όσον αφορά την οδηγία στην Ιρλανδία. Το αποτέλεσμα αυτής της αποτυχίας ορθής εφαρμογής του δικαίου είναι το ότι η βιοπικιλότητα κλίμα, δίκαιο, κράτος δικαίου, ύδατα, όλα αυτά επλήγησαν. Μιλούμε για μια περιοχή που προτεύεται το Natura 2000. Να σας πω πώς έχει το ιστορικό πλαίσιο για την εξόριση της τύρφης. Έχουμε δάφη με πάρα πολύ τύρφη στην Ιρλανδία. 20% της χώρας καλύπτεται από αυτά τα εδάφη τα οποία περιέχουν τύρφη. Βέβαια, εδώ η μετάρρυψη γίνεται για πολλούς σκοπούς. Πρώτον, έχουμε τρεις σταθμούς παραγωγής ενέργειας με τύρφη. Και είναι 3 εκατομμύρια τόνους τύρφης την, ε, τη χρονιά. Η μετάφραση γίνεται από κάποια κρατική εταιρεία, ποτέ δεν έχει γίνει όμως ε, μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον. Έχουν επιδότηση 30 εκατομμύρια από την ε, Κομισιόν σήμερα αποφασίστηκε το 2001 η οι σε αυτά τα εργοστάσια. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε την ε, τύρφη για να ζεσταθούμε και στο σπίτι. Αυτό βλάπτει τις περιοχές που από το Natura 2000. Βλέπετε εδώ αριστερά, παραδοσιακά, λένε ότι πάει ο κάποιος γερούλης με το κάρο του και φορτώνει. Δεν, είναι, δεν γίνεται έτσι πραγματικότητα. Είδαμε αυτό το παράδειγμα. Παραδοσιακό δεν είδατε όμως, δεν είδατε την πραγματικότητα που γίνεται με αυτές τις μηχανές. Και για την ε, καλλιέργεια στους κήπους και λοιπά, χρησιμοποιείται η τύρυφη, αλλά εκτός από τους ιδιώτες και από εμπόρους, όπως αυτούς που εμπορεύονται τα μανιτάρια. Εξάγουμε επίσης και στην Νότιο Αφρικανική Δημοκρατία την τύρυφη. Νότιος Αφρική προστατεύει το δικό της έδαφος και γι' αυτό ψάχνει τύρυφη από όλου. σαν να ήταν καρπός επομένως την εξορίσουμε την ε, τύρφη το 2008 ο τότε υπουργό Εμπορίου επισκέφθηκε την Νοτεφρινή Δημοκρατία και είπε ότι πρόκειται για προϊόν φιλικό στο περιβάλλον. Δεν ισχύει αυτό. Έχει τεράστια επίπτωση για την ε, αλλαγή του κλίματος, για την βιοποικιλότητα, για την ποιότητα του εδάφους. Ξέρετε ότι όταν έχουμε μέσα στο νερό τύρφη και βάζουμε τη χλωρίνη για να καθαριστεί το νερό και να το πιούμε, τότε έχουμε αποτελέσματα καρκινογόνα. Και υπάρχει τέτοιο πρόβλημα τέτοιων καρκινογόνων ουσιών στο νερό της Ισλανδίας. η, ας το πούμε, η υδροδυναμική αυτών των ε, βάλτων επηρεάζεται από αυτή την εξόριξη και γι' αυτό και έχουμε πλημμύρες οι οποίες είναι όλα πιο σοβαρές όπως είδατε πρόσφατα. Είπαμε ότι έτσι έχουμε τύρφει παντού στην χώρα και δεν λαμβάνεται υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο για τη φύση. Μιλούμε για βάλτους που βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά τη δημιουργία τους και το, η οδηγία για το φυσικό περιβάλλον τους δίνει προστασία στην προτεραιότητα μάλλον στην προστασία, συγγνώμη. Και έχουμε πάρα πολλέ πάνω από 100 τέτοιου είδους βαλτότοπους. Η οδηγία αυτή πέρασε το 92. Όμως συνεχίζεται η εξόριξη που οδηγεί σε 19 χρόνια βλάβης αλλά και εθελοντυφλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα. Βλέπετε τώρα το βάλτο Moods. Βρίσκεται στην επαρχία του Κίλτερ. Βλέπετε εδώ πόσο μεγάλη είναι η βλάβη από την εξόριξη της τύρφης. Ακόμα χειρότερα είναι τα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο. 19% αυτών των Βάλτων έχει χαθεί και βέβαια δεν έχει κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το 1 τρίτο του υπόλοιπου 1%, ε, 99% ε, ε, συγγνώμη ήταν είναι η απόλυτη, το 1% έχει γίνει τελευταία δεκαετία. Οπότε αυτό το φυσικό περιβάλλον κινδυνεύουμε το χάσουμε τα μέσα επόμενα χρόνια. πήρε τόσα χρόνια επομένω για να γίνει κάτι και αυτό το, το πρώτο διάβημα για την αφορά και τον φέτος. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Στην επαρχία του Τίπερερη βλέπετε τον βάλτο Redwood. Εδώ 85% από αυτό το βάλτο χάθηκε μεταξύ 1994 και 2005. Πήγαμε το Μάιο και μπορείτε να δείτε εδώ πώς συνεχίζεται η εξόριξη. Πήγαμε στα, σε 33 από τους 55 τέτοιους βαλτότοπους που έχουν τύρφει. Είδαμε ότι 22 είχαν ζημία, 8 από 33 ε, λαμβάνουν χρηματοδότηση για για επιδιόρθωση, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απευθύγαμε γι' αυτό σε εσά. Πιέστε. Βοηθήστε να συνεχιστεί το έργο μας. Πρέπει να αρχίσει η επανόρθωση της ζημία. Είναι επαρχιακή αυτή η δραστηριότητα. Το, την άνοιξη του γίνεται η εξόριξη, το αφήνουν να ξεραθεί και καίνεται την τύρφη των το 2012 την άνοιξη θα ξαναπάνε να εξορίξουν. Επομένω, αυτό που θέλω από εσά είναι να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να λάβει κάποια μέτρα. Παρακαλώ και η Επιτροπή σα να λάβει υπόψη αυτή την κατάσταση ότι μπορεί αυτό να είναι κάποια λύση και μιλήστε στην Κομισιόν. Έχουμε την επίσημη επιστολή του άρθρου 258. θα μπορούσε να ζητηθεί πίσω η επιδότηση. Άλλο θέμα. Η εξόριξη της τύρφης εκτός των προστατευμένων περιοχών. Βλέπετε εδώ τις περιοχές της Πορτοκαλί. Εκεί υπάρχει είναι στο περιβάλλον από την εξόριξη. Βορειοδυτικά αυτής της λίμνης δεν έχουμε προστατευόμενη περιοχή, αλλά η οδηγία για τα πουλιά προστατεύει τη λίμνη. Έχουμε εδώ βλάβη εκτός προστατευόμενης περιοχής, αλλά τελικά επηρεάζεται και η προστατευόμενη περιοχή. Εδώ βλέπετε τι έγινε επί τόπου. Δεν υπάρχει εδώ άδεια εξόριξης. Δεν έγινε μελέτη επιπτώσεων. Δεν δόθηκε έγκριση. Έχουμε απόφαση του δικαστηρίου του 1999. Η Ιρλανδία δεν αρνηθήκε ότι δεν έχει κάνει τη, τη μελέτη όπως λέει η οδηγία. Τώρα, στο τι περαίρει άλλη τοποθεσία, Και εδώ συνεχίζεται χωρίς άδεια. Η εξόρυξη δίνονται πάνω από 300.000 εκεί λέει ο μιλητής, ενίσχυση. Το 1999 είπαμε λήφθη αυτή η απόφαση του δικαστηρίου κατά δίκη της Ελλανδίας για την εξόριξη όταν πήγαμε το Μάιο. Συνεχιζόταν όμως, χωρίς άδεια η εξόριξη. Οπότε, λάβετε υπόψη την αφορά μας και κατόπιν του πρώτου διαβήματος άρχισε η Επιτροπή να ασχολείται αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η άναρχη εξόριξη εκτός προστατευμένων περιχώρων. Δεν υπήρξε άλλη απόφαση του ΔΕΚ παρά την πρώτη απόφαση. Γιατί έγινε συμβασμό. Από τότε όμως η Ιρλανδία δεν τηρεί τους όρους αυτού του συμβασμού που μπήκε για να μην πληρωθεί το πρόστιμο. Και επομένως γίνεται αυτή η δραστηριότητα παρά όλες τις οδηγίες για το περιβάλλον, ύδατα κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει επίσκεψη επιτόπου και αυτό θα ε, σας πείσει. Και μην φοβάστε θα με θεμίσει κοντά σας και δεν θα σας ρουφήξει το τέλμα, το έλος. Ε, σας ευχαριστώ για την αναφορά που παρουσιάσατε και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Λίαμ Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο αναφέρον οπωσδήποτε ευαίσθηση της προσοχή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα της Ιρλανδίας. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να δίνεται εντύπωση ότι η Κομισιόν τα τελευταία 20 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ε, ο αναφέρον έθι, ε, ε, αναφέρθηκε σε μια περίπτωση που οδήγησε σε προτινόμενα πρόστιμα για την Ελλαδία το 2005. Γνωρίζουμε το πρόβλημα της εξόρυξης ε, της τύρβης στην Ελλαδία που φτάνει μέχρι το τη δεκαετία του 90 και τότε τα μόνο μέσα που είχαμε ήταν η οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η οδηγία αυτή προέβλεπε ε, προκαταρκτική ε, αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είδαμε ότι η Ιρλανδική νομοθεσία προέβλεπε την ε, μελέτη αυτών των επιπτώσεων μόνο πάνω από πάρα πολύ σημαντικά επίπεδα. Εμείς ε, προσφύγαμε, πετύχαμε την απόφαση του δικαστηρίου το 1999 που θεώρησε ότι οι κανόνες αυτοί δεν ήταν αποτελεσματικοί όσον αφορά την οδηγία περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν είναι σωστό λοιπόν αυτή την εντύπωση του Κομισιόν δεν έκανε τίποτα. Το δεκαετία του 90 κάναμε ό,τι έπρεπε, μαζέψαμε πληροφορίες για ε, πλήγματα σε ευαίσθητες περιοχές. Τώρα, τι έγινε μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Ε, Κάνουμε ό,τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν όταν υπάρχει μια απόφαση. Πιέσαμε τους ε, υπευθυνούς να αποδείξουν ότι έχουν αλλάξει τους κανόνες για να είναι συμφωνή με το δικαστήριο. Γιατί ε, εμείς βασιστήκαμε στο ότι η εθνική νόμη δεν ήταν οι σωστοί. Όχι ότι δεν εφαρμόζεται κάτι και όταν η Ιρλανδική κυβέρνηση δεν πήρε την απαραίτητη νομοθεσία προχωρήσαμε με την επιβολή προστήμων της τάξης του 20.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος καθημερινά αλλά όταν η Ιρλανδία μας είπε ότι μπορεί να αλλάξει την νομοθεσία της ε, τώρα για να είναι σύμφωνη με, το δικαστική απόφαση ίδιος για τις ευαίσθητες περιοχές, εμείς κλείσαμε το 2005 αυτό το φάκελο. Δυστυχώς, και εδώ βέβαια συμφωνώ οπωσδήποτε με την ε, παρουσίαση των ε, αναφέροντων, αυτοί οι κανόνες δεν εφαρμόστηκαν και η νομοθεσία δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Είναι σωστό, δεν υπήρξε ποτέ αξιολόγηση των πυροβολογικών επιπτώσεων για την εξόριξη τύρβης στην Ιρλανδία. Πήραμε λοιπόν πολλές ε, πληροφορίες από τους ετούντες, αυτούς και άλλους ε, διαφερόμενους και ξανανοίξαμε μια νέα υπόθεση τον Γενάρη τρέχοντος έτος και με την προσοχή σε μια σειρά συστηματικών αποτυχιών, όπως θεωρούμε. Ε, συμφωνούμε λοιπόν με τους αναφέροντες ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση μια εφαρμογή κοινωτικού δικαίου. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρνείται η Ιρλανδική κυβέρνηση. Τι γίνεται τώρα με την προσφυγή που ξεκίνησε το Γενάρη από τη δική μας ε, σκοπιά οι πιο ευαίσθητες περιοχές είναι αυτές που ανέφερε και ο αναφέρον το 1% το 1%. Η ελληνική κυβέρνηση μας είπε ότι θα σταματήσει στις τοποθεσίες αυτές ε, η εξόριξη το 2011 στις πρώτες και ε, το επόμενο τόσο στις επόμενες. Εμείς είδαμε ότι συνεχίζεται όμως η κοπή της στήρβης, εξόριξη της και παρενεβημέν και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε ενδεχομένω τα μέτρα που είχε προβλέψει ε, νωρίτερα η Κομισιόν. Δηλαδή η κυβέρνηση είπε ότι έχει διακοπεί η εξόρυξη σε αυτές τις περιφέρειες και προωθούν ειδικά μια πολιτική διακοπή τη κοπή τύρφης. Σταματήστε δηλαδή σε αυτές τις ε, κεντρικές ε, περιοχές και εξετάζουμε πώς εφαρμόζονται οι κανόνες για γενικά τις ε, περιοχές που έχουν τύρφη, όχι μόνο τις ιδιαίτερα προστατευόμενες και η Ιρλανδική κυβέρνηση μας είπε ότι θα μας υποβάλει κάποιες προτάσεις και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι θα προωθήσουμε την δικαστική προσφυγή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποδεκτικά στοιχεία που μας δώσατε αναφέροντας και νομίζω ότι αυτή μας η απειλή είχε ήδη επιπτώσει σήμερα. Ευχαριστώ η κυρία Άουκεν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες είναι από τα χειρότερα που έχουμε δει. Φαινόταν ότι οι αρχές ίσως να έδιναν υποσχέσεις αλλά δεν κάνουν τίποτα. Σαν να μην φοβούνται τίποτα επίσης. Ότι μπορεί να συνεχιστεί. Παλιά υπόθεση που παραβιάζει όλους τους κανόνες. Το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκάθαρα. σαν να είναι στη σελήνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο συμβαίνουν στην Ιρλανδία δεν ανησυχούν κανέναν. Εκτός. Χαιρόμαστε που φέρατε εδώ την υπόθεση. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η απάντηση τώρα που το θέσατε το θέμα στην κυβέρνηση. Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας δεν πρέπει να είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Πάντα στο Κοινοβούλιο τη Δανία συζητούνται τέτοιες υποθέσεις. Προσπαθήσατε να προσφύγετε στο δικαστήριο στην Ιρλανδία. Πρέπει να χρησιμοποιούμε και τι εθνικές δυνατότητες. Υπάρχει παράβαση του νόμου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τίποτα δεν συμβαίνει η αλληλογραφία, η λογογραφία αλλά τίποτα. Υποστηρίζω τους αναφέροντες. Εάν υπάρχει δυνατότητα να αναλυφθεί η δράση, τώρα πρέπει να γίνει. Διότι γίνεται αυσιολογή τύρφης και στη Δανία. Πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να βοηθήσουμε με τους, αυτούς που καλλιεργούν τους κήπους τους με λιπάσματα. Συνδέεται και με τα πόλη, το συζητούσαμε πριν. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Αντί να προξενούμε βλάβες, μπορούμε να βρούμε επικοδομητικές λύσεις. Σαφή διατύπωση χρησιμοποίησατε. Περιμένω όμως μια πιο ξεκάθαρη απάντηση όσον αφορά τη συνέπεια στον αντίκτυπο που έχει αυτή η εξόριξη τύρφης για το περιβάλλον. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, first of all, I want to... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των προστατευόμενων περιεχών και εκείνων που δεν είναι. Και επίσης συμφωνώ με τον Πρόεδρε ότι εκτός προστατευμένων περιεχών η νομοθεσία για την αξιολόγηση ε, κατεπατήθη. Υπήρχε, αλλά δεν την τήρησαν. Τώρα έχουμε πάντως τη σχετική νομοθεσία, η είναι και μάλιστα αυστηρότερη όσον αφορά αυτό. Οπότε συμφωνώ με αυτά που είπατε και στις προστατευμένες περιοχές τα πράγματα αλλάζουν εντελώ και εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι διαφορετικό ε, και να σας δώσω μια άλλη εικόνα. Πρώτα πρώτα είναι πάρα πολύ σημαντικό το, το ότι είπε η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να σταματήσει η εξωτική δραστηριότητα. Και όποιο συνεχίσει να το κάνει αυτό, παρανομία. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να λάβουμε υπόψη ότι συνεχίζεται η δραστηριότητα αυτή και από φυσικά πρόσωπα, όχι από εταιρείε, γιατί οι γονεί και, και προ πάβο κάνουν αυτή τη δραστηριότητα. Επομένω, ζητείται από κάποιου Ευρωπαίου να απεμπολίσουν κάποια του δικαιώματα και αυτό το οποίο τώρα προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να θεσπίσει μια δέσμη μέτρων είτε για αντιστάθμιση να δίνει κάποια χρήματα εταιρείως ή να τους δίνει κάποια άλλα καύσιμα τα οποία τα, ε, σε σχέση με αυτήν την ε, να φύγουν τέλο πάντων από την, από την τύρφη και να πάνε αλλού ή να πάνε τουλάχιστον σε μέρο που δεν προστατεύεται. Ε, Κάναμε μια συνάντηση με 40 τέτοιους ε, χρήστες και εξορίκτες και τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο ε, απλά όπως τα λένε οι αναφερόμενοι. Εγώ μίλησα με κάποιον ε, την Πέμπτη. Αυτός έχει 17 εκτάρια τέτοιου βάλτου και είπε 16,5 εκτάρια σας τα δίνω. Θέλω όμως μισό εκτάριο από αυτό το βάλτο όπου μπορώ εγώ και τα παιδιά μου να κάνουν αυτό που κάνουν, κάνουμε πάπο προς πάπο. Ε, Επομένω, τι να του πω, δεν μπορούσα να του πω τίποτα, να τον, δεν μπορούσα να, τον ε, παρηγορήσω για αυτό το οποίο ζητούσα, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει ε, κάποιο τέτοιο πακέτο με αποζημίωση. 15 χρόνια γίνεται αυτό, αυτή η προσπάθεια, αυτή η εξορρυκτική. 250.000 ευρώ κοστίζει ένα τέτοιο εκτάριο, αλλά το ζητάμε κάτι να κάνουμε χωρίς να δίνουμε την αντιστάθμιση. Επομένως η παρουσίαση είναι ενδιαφέρον να αναλάβει την υπόψη ότι το επόμενο θέμα της κυρίας Βαλέαν αφορά δικαιώματα πολιτών. Γιατί έχουμε χιλιάδες Ιρλανδών που δικαιούνται την εξόρυξη και θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους αφαιρεί αυτά τα δικαιώματα και δεν τους δίνει τίποτα σε αντιστάθμιση. Επομένως, έχω πω το εξή. Δεν θέλουμε αντιστάθμιση και αντιπαράθεση. Θέλουμε συνεργασία. Και νομίζω ότι ω επιτοπλίστων είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα. Ναι, ωφελεί να επισκεφτείτε επιτόπου, αλλά εκτό από τα χωράφια, επισκεφτείτε και τον κόσμο αυτού που επί αιώνες κάνουν την εξόριξη στα ίδια αυτά μέρη και πασχίζουν και αυτοί να βρουν μια λύση που να είναι εφαρμόσιμη. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος αισθάνεται θυμό και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ. Δεκάδες χιλιάδων στην Ιρλανδία υπογράφουν αναφορές που θα σας τις στείλουν. Γιατί θεωρούν ότι τους μπλοκάρετε από μια πάρα πολύ μακριώνα παράδειση. Συμφωνώ σε πολλά πόσα όσα είπαν οι αναφερόμενοι. Όμως, Υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα που δικαιούνται να εξορίσουν την τύρφη και για αυτού θα πρέπει να βρούμε κάποιε λύσει. Άρα χρειάζεται συνεργασία. Όχι αντιπαράθεση. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή σα Όλα αυτά να τα λάβει υπόψη. Αυτό Θα δούμε στο επόμενο θέμα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν εδώ λύσεις ευρωπαϊκές, όπως έχουν παράδοση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. E, ε, Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Χάκιν. Γιατί όλοι γνωρίζουν ε, τώρα πια πόσο συναισθηματικά φορτισμένο είναι το θέμα αυτό στην Ολλανδία και πολιτικά. Και η σημερινή κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το τόσο ακαθόδες πρόβλημα που ε, κληρονομήθηκε γιατί από το 97 έχει αγνοηθεί τελείως το θέμα ε, λες και πρόκειται να εξαφανιστεί από μόνο του. Τούτου λεχθένως όπως σας είπα, είναι συστηματικά φορτισμένο το θέμα και πολλοί είναι ιδιαίτερα προσκολλημένοι στην περισυλλογή της τύρφης, στην εξόριξη της ε, Τη Βέβαια υπάρχουν βλάβες. Χρειαζόμαστε νομίζω τη βοήθεια της Κομισιόν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο να βρεθεί η λύση διαπραγματευτικά. Και θα ήταν χρήσιμο παραδείγματο χάρη του χρόνου να υπάρχει μια επιτόπου επίσκεψη υπαλλήλων της Κομισιόν αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αγνοούμε την γενική εικόνα, όχι μόνο τι προστατευμένε περιοχέ. και παρακαλώ την Κομισιό να ανταποκριθεί στο αίτημα των ε, mm. κ. Ζηγιά. Mm. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που με ενοχλεί κάπως είναι ότι καμιά φορά και τα κράτη-μέλη μια λένε έτσι και μια λένε αλλιώ. Δηλαδή το Natura 2000 δεν ήρθε εξ ουρανού. Τα κράτη-μέλη συμμετείχαν ενεργά για να προετοιμάσουν σχετική νομοθεσία. Τώρα πάνε ε, πίσω στις πατρίδες μετά που θα έχουν πάρει την απόφαση στις ε, Βρυξέλλες και όταν φτάσουν στο σπίτι ξεχνάνε τι είχαν αποφασίσει στην, ε, στις Βρυξέλλες. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν άμεσα διαφερομένοι, ότι όταν υπάρχει παρέμβαση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας ε, πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσεις. Τώρα να δοθεί εντύπωση ότι όλα αυτά ξαφνικά εξ ουρανού εμφανίστηκαν και ότι φταίει οι Βρυξέλλες, φταίνουν, φταίνε, δεν νομίζω ότι είναι πολύ τίμιο. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα αυτό αγνοήθηκε για χρόνια και χρόνια. Δεν ξέρω, φαντάστηκαν ότι θα το λύσει ο Θεούλης το πρόβλημα αλλά δεν το λύνει. Μεγάλωσε. Και τώρα είδαμε ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται εξορροστήρυφη στις προστατευόμενες περιοχές. Ναι, αυτό ήταν κάτι που το ξέρανε όμως από πολύ καιρό. Τώρα δεν επιτρέπεται λοιπόν να κάνουμε τους ιδιοκτήτες να επαναστατήσουν κατά της Ευρώπης. Όχι, πιστεύω και εγώ θα πρέπει λίγο να έχουμε ένα διάλογο. Καταλαβαίνω και τους ιδιοκτήτες. Πρέπει να το εξηγήσουμε ε, αλλά βέβαια υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί. Αλλά είπα και χθε ότι συγχύζομαι με τα κράτη-μέλη. Αποφασίζουν κάτι στι Βρυξέλλε, πάνε πίσω και ξεχνάνε τι έχουν αποφασίσει. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Γιατί έτσι καταστρέφουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο. Natura 2000 είναι περιφέρειες προστατευόμενες και υπάρχουν λόγοι για κάτι τέτοιο και θα πρέπει να εφαρμοστεί λοιπόν η νομοθεσία. Μία ερώτηση προς τους αναφέροντες. Εγώ θέλω να μείνει ανοιχτό, να υπάρχει ένας διάλογος και με την ελληνική κυβέρνηση, έντονος διάλογος όσον αφορά και αποζημιώσεις. Η μόνη ερώτηση που έχω προς τους αναφέροντες γιατί είπε η Κομισιόν ότι κάτι βελτιώθηκε. Εσείς ε, πραγματικά είδατε στι προστατευόμενε περιοχέ να υπάρχει κάποια θετική κίνηση. Yes. Thank you for the questions. Uh, perhaps... Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να απαντήσω με τη σειρά. Κάτι γενικό. να τονίσουμε ότι πολλές συζητήσει εστιάζονται επί των προστατευμένων τοποθεσιών Natura 2000. Είναι σημαντικό να τονίσουμε και οι μη καθορισμένες περιοχές τι γίνεται. Αυτό το θέμα εκείνων που συλλέγουν την τύφη e είναι σημαντικό. Θεωρούνται ότι είναι θύματα, θεωρούνται σε αυτούς τους θύματα. Θεωρούνται ότι καλύπτονται οι περιοχές Natura 2000 ενώ οι μεγάλες εταιρείες κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενική. Όχι μόνο Natura 2000. Τι γίνεται με τις μεγάλες επιχειρήσεις. ως συγκεκριμένα τώρα. Αυτά που είπε και ο Σκάσμαν. Είπε ότι είπαμε κάτι λάθος και ότι κινήθηκε την τελευταία 20 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ τι είπα. Ήταν 20 χρόνια, 19 χρόνια από την οδηγία ε, του 1992, του Habitat. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2001 δεν είχε κάνει τίποτα. Η οδηγία EIA ήταν η νομική δράση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φορούσε την Ιρλανδία όλοι. Καλή δράση για Natura 2000, για τις περιοχές Natura 2000. Όσον αφορά τι μη καθορισμένε περιοχέ και τη νομική μα δράση, που την ξεκινήσαμε, την κλείσαμε και ανοίξαμε νέα υπόθεση, δεν ήταν ξανοίξαν την παλιά υπόθεση. Θα ήταν η οδηγία EIA. Αλλά ξεκίνησε νέα υπόθεση για την Natura 2000. Δεν έχουμε πλήρη νομική κάλυψη στην Ιρλανδία. Θα συμφωνεί και ο κ. Κάσμαν. Η κυρία Άουκεν. Χαιρόμαστε που αναγνωρίζει ότι είναι από τις χειρότερες υποθέσεις που έχει εξετάσει η Επιτροπή. Διάλογος εκτός μικροφώνου, δεξί κυρία Άουκεν και το αναφέροντος. Τι κάναμε σε εθνικό επίπεδο ήταν η ερώτηση. Προσπαθήσαμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο το 2002. Για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις πρόβλημα μεγάλο στην Ιρλανδία είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Το νομικό κόστος μπορεί να φτάσει εξαψήφια στοιχεία, πάνω από 100.000 ευρώ για νομική δράση. Και νομικοί μας είπαν ότι δεν βγαίνουμε πουθενά έτσι. Φοβηθήκαμε τη χρεοκοπία. Πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει για το περιβάλλον εργάζονται βάσει εθελοντών και ο Ντέιβιτ και εγώ είμαστε εθελοντέ. Χάρκιν. Αναφέρθηκε στην κληρονομιά τη συλλογή τύρφης η φυσική κληρονομιά της Ιρλανδίας ανήκει στους αγέννητους Ιρλανδούς. Δεν ανήκει σε ελάχιστους αυτούς που μαζεύουν την τύρφη. Ανήκει σε όλους. Χρειαζόμαστε λύση. Θα υπάρξει σύγκρουση την άνοιξη, είναι σίγουρο. Τσόλτερς έκανε καλά σχόλια. Γιάρ, αν βελτιώθηκαν οι τοποθεσίες Natura 2000, όχι. Τον Μάιο 2011 επισκεφτήκαμε τις περιοχές. Μετά ακολούθησε η ανακοίνωση τον Ιούνιο σταμάτησε η συλλογή τύρφης τον Ιούνιο, έτσι κι αλλιώς σταματάει η συλλογή, σταματάει τον Ιούνιο, αυτή την εποχή αφήνεται να στεγνωθεί. Την άνοιξη του 2012 το θέμα τι θα γίνει. Θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, πρέπει να απαντήσουμε σε, σε κάποιες ερωτήσεις. Στις 12.30, σε λιγότερο από 20 λεπτά, λέει η Πρόεδρος, πρέπει να φύγουν οι διερμηνείς. Μπορούμε να αλλάξουμε κάπως το πρόγραμμα, την ημερήσια διάταξη και να πάμε στο θέμα 2 το θέμα 23 και να αφήσουμε την έκθεση Βάλιαν να την κάνουμε μόνο στα αγγλικά, χωρίς διερμηνής. Συμφωνούν τα μέλη. Πάμε στην παρουσίαση λοιπόν της υποθέσεως του σημείου 23. Είναι εδώ οι αναφέροντες νομίζω.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 καθώς περιμένουμε την εγκατάσταση